Okay. On va commencer. Πρόεδρος, ξεκινούμε. Καλημέρα σε όλους και συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση. Γίνονται κάποιες μικρές διορθωτικές ε, κινήσεις τεχνικού χαρακτήρα για κάποιες συνδέσεις. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Το πρώτο θέμα είναι έγκριση μερικές διατάξεις. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι πάνω σε αυτό. Εάν ναι, τότε πάμε στο 2. σημείο 2 το οποίο είναι οι ανακοινώσει ε, της Προέδρου. Έχουμε τρία κατεπήγοντα ψηφίσματα ε, κατά την Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Πρώτα-πρώτα όσον αφορά τα πρόσωπα ΛΟΑΔΚΙ στην Ουγκάντα, τον ποινικό κώδικα της Ινδονησίας και τρίτον Αίγυπτος. Και τα τρία μας απασχολούν. Ε, σοβαρά προβληματιζόμαστε σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οπότε θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, να δοθεί συνέχεια εδώ στην ε, Υποεπιτροπή Ανθρωπινών Δικαιωμάτων, να δούμε τι θα γίνει, πώς αυτά τα κατεπήγοντα ψηφίσματα ε, θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή μας στο μέλλον. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι από αυτού. Οπότε πάμε στο 3. Έγκριση των πρακτικών των ε, συναντήσεων 25 και 26 Σεπτεμβρίου και 8 Οκτωβρίου. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, τότε τα πρακτικά εγκρίνονται. Και τώρα, τέσσερα. Ανταλλαγή απόψεων με γυναίκες που υπερασπίζονται τα περιβαλλοντικά και γεωκτητικά δικαιώματα και δικαιώματα των αυτοχθόνων στην Λατινική Αμερική. Έχουμε εδώ εκπροσώπους ε, Κολομβίας, Ουνδούρας, Γουατεμάλας και Μεξικού. Είναι σημαντικό να ε, εξετάσουν το θέμα αυτό των περιβαλλοντικών και δικαιωμάτων ε, από πλευράς γυναικών. Ε, αυτό η έλευσή σας εδώ για μένα κάτι πολύ ευχάριστο και αναλάβαμε εδώ στην Επιτροπή μας να μπορέσουμε συστηματικά να παρακολουθήσουμε τα ζητήματα αυτά που είναι μια προτεραιότητα για την ε, Υποπιτροπή μας. Και επίσης σε σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών, αυτά μας ε, απασχολεί γιατί πρόκειται για τμήμα του πληθυσμού πιο ευάλωτο για αυτά τα ζητήματα, αλλά επίση να δούμε και πώς είναι δυνατόν να είναι παράγοντες ε, αλλαγής οι γυναίκες. Οπότε δεν λέμε μόνο για τις ε, γυναίκες ως θύματα, αλλά τις γυναίκες ως φορείς αλλαγής. Οπότε αυτό θέλουμε να δούμε στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα, θα δώσουμε τώρα το λόγο ε, στις ε, φιλοξενούμενές μας, που ξεκινούμε την κυρία Φρανθέσκα Νούνιες. Η προσωπή της Διεθνής Ταξιαρχίας Ειρήνης. Κατόπιν κυρία Σάντρα Καλέλ, ε, εκπροσωπή, τους Μάγια ή την Μάγια από την Γουατεμάλα, ε, την, τον φορέα οργανώσεις Βαραπασένσε, κατόπιν η κυρία Νόρα Ραμύρες από το Κέντρο Αγροτών Εργατών της Γης, κυρία Βεντάνιο, στη συνέχεια που ε, είναι και αυτή από τις ταξιαρχίες Ειρήνης, που ε, εκπρόσωπη στη κυρία Έμιλη ε, Γούλφ, από το Consortium αξάκα. Και τώρα, Όλγα Αραούχα, Έρευνα και κοινωνική δράση. Φραντσέσκα Νούνιας πρώτη, για πέντε λεπτά. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτα-πρώτα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε για μας είναι πολύ σημαντική η επιτροπή σας για να υπάρξει ε, ένας διάλογος, να καταλήξουμε σε κάποιες εγγύησει για τις ε, γυναίκες που αγορίζονται για δικαιώματα, ε, για το περιβάλλον στις χώρες μας, Κολομβία, Ανδούρα, Γουατεμάλα και επίσης στις 7 Νοεμβρίου κάναμε μια κοινή ανακοίνωση ε, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ε, από πλευρά Ηνωμένων Εθνών και εκεί είπαμε επακριβώς ότι εκφράζουμε την ανησυχία μας για το ότι συνεχίζονται τα φαινόμενα της επιδείνωσης όσον αφορά ε, την εγκληματικότητα κατά των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αμερική. Και έχουμε εκεί, αναφέρουμε διάφορα θέματα που αφορούν την ε, Κολομβία που είναι η πιο επικίνδυνη ε, χώρα για, τις, ε, για τους ακτιβιστές αλλά και η Ονδουρέ, αλλά και το Μέξικο. Και επισύρτη προσοχή στο ότι κινδυνεύουν αυτοί οι οποίοι παλεύουν για τα γεωκτικά δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά. Ε, Επίσης, στο 2018 κάνατε ένα ψήφισμα πολύ σημαντικό για την ισότητα των δύο φύλων και το περιβάλλον και ακριβώς αναφέρονται ότι υπάρχουν κίνδυνοι και για άντρες και για γυναίκες ε, ακτιβιστές αλλά οι γυναίκες ε, υποφέρουν και από σεξουαλική βία, απειλές για την οικογένειά τους, από σεξισμό, ε, υφίστανται σωματική βία, βασανιστήρια. Ε, υπάρχει κάποιος πατριαρχή βία σε σχέση με τον ρόλο της γυναίκας στο, στην κοινωνία, σε σχέση με την κατάληψη των παραδοσιακών τους ε, ε, ρόλων. Αυτό αφορά λοιπόν τους αυτόχθονες και υφίστανται δεσμενής διακρίσεις και περιθωριοποίηση. Πριν δώσω τώρα στις συντρόφισσες από τις άλλες χώρες την σκητάλη, θέλουμε να σας πούμε ότι στις χώρες μας. Ε, προσπαθούμε να συνασπίσουμε κόσμο για ε, τη, τους σκοπούς μας, έχουν πολλές επιθέσεις, ε, έχουμε δολοφονίες για ακτιβιστές, αλλά όμως υπάρχει ταυτόχρονα και ατιμορρησία. οπότε θα πρέπει να, να φωτιστούν, να πέσει φως, δηλαδή να λυθούν αυτά τα εγκλήματα και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους δολοφόνους. Πολλές φορές είναι κάποιοι πληρωμένοι δολοφόνοι. Ε, και πολλές φορές όμως υπάρχει και κάποιο είδους διαπλοκή ε, με τις αρχές της χώρας. Αυτό επομένως συνεχίζεται και αυτό δεν διευκολύνει τα πράγματα, άρα θα πρέπει να υπάρξουν εγγύησεις ότι δεν θα υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Επίση, οι ακτιβίστριε υποφέρουν κυρίω όταν είναι στην ε, Ήπεθρο, πιο απομονωμένε, δεν έχουν ε, καν πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Άρα και αυτέ θα πρέπει να βοηθήσουμε στον αγώνα του. Επίση, πάρα πολλέ αυτέ τι επιθέσει ε, γίνονται στην Ήπεθρο, γίνονται στην περιφέρεια κάποιων πόλεων, εκεί που επίσης όπου έχουμε κάποια μεγάλα έργα, μεγάλα έργα βιομηχανικά, υποδομών, ε, τουρισμού και γίνονται αυτά τα μεγάλα έργα χωρίς να εμπλέκονται οι κοινότητες που φύγονται από αυτά τα μεγάλα έργα. Οπότε πολλές φορές ε, αυτά γίνονται και με βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή πολλές φορές γίνεται ε, όλο αυτό για να παραχθούν κάποια προϊόντα που μετέρχονται στις αγορές της Ευρώπης. Και πολλές φορές έχουμε ομάδες ενόπλων ε, που δρούν σε κάποιες περιοχές που έχουν ε, πλούσιους πόρους, που είναι πλούσιες, όλα αυτά γίνονται χωρίς να εμπλέκεται το κράτος και ο στρατός. Εμείς δεχόμαστε πάρα πολλές καταγγελίες για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλους αυτούς ε, και από τις παράνομες αυτές ένοπλες ομάδες και από τη σκήτα στη Χάιβδη πηγαίνουν εκεί οι γυναίκες γιατί μια ομάδα αντίπαλη της άλλης ε, της κατηγορεί γιατί πήραν το μέρος των αντιπάλων. Και αυτά γίνεται όσον αφορά τη βία, αλλά επίσης έχουμε αύξηση ε, της εγκληματικότητα, ε, εις βάρος των ακτιβιστών. Πολύ βία που γίνεται και κυρίως με αφορμή τις ε, κοινωνικές διεκδικήσεις που πολλές φορές ε, γίνονται ε, κόντρα σε αυτά τα πολύ μεγάλα έργα. Γίνεται όπως είπαμε από τις κοινότητες που θίγονται, γιατί αυτές οι κοινότητες από τα έργα αυτά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο νερό ή σε άλλους φυσικούς πόρους. Είμαστε σε, στην πρώτη γραμμή ε, και γι' αυτό ακριβώς και είμαστε ο στόχος των εγκληματιών. Ε, επίσης, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό ότι υπάρχουν εκστρατείες δυσφήμισης και επίσης ε, γίνεται και χρήση της δικαιοσύνης ούτως ώστε αυτές οι γυναίκες ακτιβίστριες να δικάζονται και να φυλακίζονται, στιγματίζονται. Ε, έχουμε αυτή τη λεγόμενη ιδεολογία του φίλου, του διαφορετικού φίλου. Αυτά γίνονται παντού στην Νότια Αμερική. Ε, λένε ότι ε, για όλα αυτά είναι θέμα φεμινισμού, θέμα των γυναικών ακτιβιστριών ε, για πολιτικοποίηση των γυναικών και ε, τελικά κατηγορούνται αυτές οι γυναίκες ως ε, τρομοκράτησες που απλώς θέλουν να προστατεύσουν τον τόπο τους. Λένε ότι εμπλέκονται και με παράνομες ενόπλες ομάδες. Οπότε κατηγορούνται για τρομοκρατία και φυλακίζονται. Αυτό φυσικά είναι απόπειρα θύμασής τους. Και επίσης θίγονται οι φορείς τους και οι οικογένειές τους από όλα αυτά. Επίσης δεν υπάρχουν κρατικά προγράμματα προστασίας, υπάρχουν και νεανέπαρκοι, ε, υπάρχουν και πρόβλημα όσον αφορά τους μισθούς και δεν εφαρμόζονται αυτά που προβλέπει ο νόμος όσον αφορά άντρες και γυναίκες παρά το ότι η ισότητα προβλέπεται και νομοθετικά. Αυτά γιατί ξύνησα το χρόνο μου και σας ευχαριστώ. και Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα, για να δώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο χρόνο σε εσά τις παρουσιάσεις, ε, να μην ρωτήσει κανείς τώρα τίποτα, αλλά μετά. Ε, να έχετε τόσο χρόνο μπορείτε. Και τώρα, κυρία Σάντρα Καλέλα. Eh, Καλησπέρα λέει κυρία Καλέλ. Ονομάζομαι Σάντρα και προέρχομαι από την Γουατεμάλα, από την βόρεια περιοχή της ε, χώρας και συμμετέχω σε μια οργάνωση βάσης. Ε, μια οργάνωση που αφορά ε, τον κόσμο της υπαίθρου και είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ κοντά σας για ένα... Ε, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι μάγια από Κοντσί, είμαι αυτόχθον και προέρχομαι από, τέτοιες, μια τέτοια κοινότητα ε, εκεί που έχουμε αναπτύξει αγώνες αντίστασης και έτσι και συνειδητοποιήσαμε το τι γίνεται, ε, τι υποφέρουμε, μας διώχνουν από την πατρίδα μας, από τη γη μας και επίσης υποφέρουμε από την ε, εγκληματικότητα. Επομένω, ε, υφιστάμεθα τριπλές επιθέσεις ε, ως γυναίκες, ως αυτόχθονες, αλλά και επειδή είμαστε αναλφάβητοι. Και όλα αυτά μας έχουν στριμώξει. Είναι δύσκολη η κατάσταση για μας ως γυναίκες και ε, γι' αυτό ήρθαμε σε εσάς και σας είμαστε ευγνώμες, μας δίνετε αυτή την ευκαιρία και στη χώρα μας. Έχουν αυξηθεί δολοφονίες, η εγκληματικότητα, η δίωξη με φυλακίσεις των ηγετών μας και επομένως διαπιστώνουμε ότι ο πρόεδρος μας στην Γουατεμάλα Μα έχει οδηγήσει αντί να μα προστατεύσει σε μια κατάσταση πολιορκία. στρατιωτικοποίηση υπάρχει ε, στις πόλεις και στα χωριά, οπότε κάτσαμε και αναλύσαμε τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση πολιορκία. Εγώ προέρχομαι από ένα δήμο, μια κοινότητα, εκεί που υπάρχει πρόβλημα ε, ε, έχουμε δραστηριότητες υδροελεκτρικές και εξορρυκτικέ. Ε, όλα αυτά οδήγησαν στο να μας ε, κατηγορήσουν, να μας θεωρήσουν εγκληματίες εμάς που υπερασπιζόμαστε τη γη μας και επίσης υπερασπιζόμαστε το περιβάλλον μας. Ε, υπάρχει μεγάλος φυσικός πλούτος από αυτά τα φυσικά δάση. Ως ε, αυτόχθονας εμείς αντιστακόμαστε. Αντιστακόμαστε για να προστατεύσουμε τη γη μας και το περιβάλλον που το έχουμε εμείς και δεν το έχουν άλλοι οπότε το θέμα είναι ότι δίνουμε και τη ζωή μας γι' αυτό. Είχαμε μάρτυρες σε όλους αυτούς τους αγώνες. Όλα αυτά είναι πολύ οδυνηρά σε μας ως λαό. Και ήρθαμε εδώ, σε αυτόν τον χώρο, σε αυτό το βήμα που μπορούμε να σας τα πούμε. Και εσείς όμως με τη σειρά σας να πάτε να τα πείτε σε κάθε χώρα. γιατί αντιστεκόμαστε και δίνουμε αυτούς τους αγώνες, αλλά το θέμα είναι ε, από εδώ, από τη δική σας θέση κάτι να κάνετε να αλλάξουν οι πολιτικές. Γιατί αναλύθηκε από εμά το πώς μπορούμε να έχουμε κάποια ανάπτυξη, αλλά να υπάρχει κάποια διαβούλευση πριν τα έργα, πριν την ανάπτυξη, να είναι σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και είπαμε ότι θα πρέπει κανείς επιτόπου να πηγαίνει και να διαπιστώνει πώς ζούμε εκεί στις πόλεις και στα χωριά μας γιατί όλα το είναι απλώς ασκήσεις επί χάρτου όσα γίνονται, όσα κουβεντιάζουν οι πρόεδροι των χωρών. Εκεί όμως, επιτόπου να πάει κανείς να δει τι κατάσταση επικρατεί και τι τραβάμε ως λαός. Οπότε γι' αυτό ήρθαμε να σας τα πούμε, ε, θέλουμε να κάνουμε και κάποια παρουσίαση, αλλά δεν γίνεται για να σας δείξουμε ακριβώς τι υποφέρουμε στις πόλεις και στα χωριά μας. Οπότε, στην βόρεια περιοχή της χώρας υπάρχει ένα φαινόμενο πιο έντονο. Εκεί υπάρχει, είπαμε, φυσικός πλούτος και εκεί δίνουμε τον αγώνα. Ε, πριν από δύο μήνες ξεκίνησε αυτή η κατάσταση πολιορκίας σε πόλεις και χωριά και υπήρξε και ένοπλη σύγκρουση. Οπότε φοβόμαστε ότι θα έρθει ο στρατός. Και όλα αυτά γιατί θέλουν να εκμεταλλευτούν τον πλούτο της περιοχής μας. Και αυτό θέλουμε να σας ε, ζητήσουμε ως λαός, ως χώρα, ως περιοχή, ότι θα πρέπει αυτά να τα δείτε γιατί αυτό αφορά πολλές χώρες, γιατί πολλές χώρες έρχονται να εκμεταλλευτούν το φυσικό πλούτο μας. Όμως θέλουμε να ζητήσουμε το εξή. Θα πρέπει να ερωτάτε ε, πρώτα ο ενεχόμενος λαός, ο φυγόμενος κάθε φορά λαός. Γιατί ε, υπάρχει καταπάτηση των, δικαιωμάτων μας ως γυναικών. Αυτό είναι το δίνηρο. Και επίσης εδώ θα πρέπει εσείς από αυτή τη θέση να παρακολουθήσετε τις εξελίξεις, να δείτε τι μπορεί να γίνει με το ψήφισμα του 2018, εκεί που θίγεται το πρόβλημα των γυναικών. Αυτό θέλουμε να σας πούμε. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το θέμα. Αυτό θέλουμε να σας ζητήσουμε. Γιατί υπάρχει αυτό, αυτή η συμφωνία, υπάρχει αυτό το ψήφισμα, αλλά θα πρέπει να λάβει σάρκα και ώστα και αυτό μας απασχολεί και αυτό ήρθαμε να σας εξηγήσουμε εδώ, σε εσά εδώ, σε εσά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ευχαριστούμε. Ε, και εμείς ευχαριστούμε, λέει κυρία ε, Αρενά. Και τώρα η κυρία Ραμύρες από την Ονδούρα. Γεια σας και καλησπέρα. Νόρα Ραμύρες ονομάζομαι και ανήκω σε κάποια οργάνωση οποία αφορά τους εργαζόμενους στην Ήπεθρο σε αγροτικές εργασίες. Το 85 ιδρύθηκε η οργάνωσή μας, αλλά εδώ και τρεις αιώνες αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα των γεωργών, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την περιοχή μας, για την κοινή κληρονομιά, περιουσία. Και πάντα όπως ε, είπε η συντρόφισσα, έχουμε ένα σωρό προβλήματα. Όπως είπαμε, υφιστάμεθα πάρα πολλά εγκλήματα, την εγκληματικότητα ε, των ε, φεουδαρχών και από πλευράς κρατικής. Οπότε τώρα το πρόβλημα είναι το εξής. Έχουμε 6.000 ε, γεωργούς, 30% γυναίκες που υποφέρουν, που ποινικοποιείται η δράση τους. Και το πράγμα που το κακό στο χειρότερο και μεταξύ άλλων θα πρέπει να παλέψουμε. Θα πρέπει να κατεβούμε στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο. Όμως ποινικοποιείται η δράση μας. Δεν μπορούμε να κατέβουμε στο πεζοδρομείο, διότι μας κατηγορούν. Λένε ότι δήθεν είμαστε τρομοκράτες. Βία, απειλές κατά των οικογενειών μας. Μας λιθοβολούν, έρχονται και πολιορκούν τα γραφεία της οργάνωσης. Χρησιμοποιούν και το στρατό. και βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλοί οι ε, συμπατριώτες που παραπέμπονται στη δικαιοσύνη. Στην Ονδούρα και αλλού. Απειλές. Οπότε με θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να ληφθεί πως αυτό αφορά πολλές οργανώσεις θα πρέπει να δοθεί βοήθεια τελικά πολλές οργανώσεις βοηθούν προσπαθούν να βοηθήσουν αλλά δεν φτάνει αυτή η βοήθεια στον κόσμο δεν φτάνει σε δήμους και κοινότητες ζούμε υπό απειλή. Οι περισσότερες από αυτές τις φυγόμενες γυναίκες από εμά που αγωνιζόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα ημών των γυναικών, μας μπλοκάρουν. Λένε ότι όλα αυτά απαγορεύονται Και έτσι η δράση μας δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και είμαστε σε πολύ αδύναμη θέση. Οπότε έχουμε φτάσει στα όρια μας ως γυναίκες ακτιβίστρες. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε λόγω αυτών των απειλών αυτής της ποινικοποίηση. Πολλέ γυναίκες εγκαταλείπουν το σπίτι τους, τι οικογένειε, τη χώρα. Λόγω των αγώνων που δίνουν για τη γη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε όλοι να μπορούν να ζήσουν στην χώρα μας, αλλά δυστυχώς το 60% της γης μας έχει παραχωρηθεί σε Αμερικανούς και άλλους. Αυτοί αρπάζουν τον πλούτο της γης μας. Πρόεδρος. Ευχαριστώ όλοι Και τώρα. Κύριε Από το Μεξικό. Ευχαριστώ πολύ. Η Emily De Wolf από το consortium ο Αξάκα δεν μπόρεσε να έρθει. Αλλά θα μιλήσω εγώ για, στη θέση της. Ε, στην πολιτεία ο Αξάκα είναι η δεύτερη πιο μεγάλη πόλη και περιοχή ε, όπου έχουμε επιθέσεις ε, σε αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να αγωνιστούν για το περιβάλλον. Είναι λοιπόν το δεύτερο μέρος το πιο περιβάλλον, ε, το πιο πιθανό για τις ακτιβίστριες. Φέτος είχαμε πέντε τέτοιους ακτιβίστριες, ακτιβιστές που ε, ειχαν εκεί, τέσσερις από αυτούς ήταν για τα ανθρώπινα δικαιώματα των αυτοχθόνων. Και η βασική τάση που αφορά τις γυναίκες ακτιβίστριες, για το Consortium Αξάκα και άλλες οργανώσεις είχαμε τρεις διαφορετικές τάσεις, ακριβώς αυτά τα οποία είπε η κυρία ε, η συντρόφισσα Νούνια στην εισαγωγή. Επίσης, ε, βλέπουμε ότι έχουμε δύο κατά των γυναικών και έχουμε κάποια στοιχεία του consortium που όλα αυτά τα έχουν καταγράψει και 2010-2016 527 ε, δολοφονίες γυναικών και μόνο το τελευταίο χρόνο ε, πάνω από 300 γυναίκες δολοφονήθηκαν και ε, οπότε συνεχίζεται αυτή η των γυναικών και τα μέτρα τα οποία λήφθησαν δεν ήταν επαρκή για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα μπορούσαμε επίσης να αναφέρουμε τη Μαρία Δελσόλ Κρούθ Χαρκίν. Αυτή ήταν ε, στις 2 Ιουνίου του 2018, έπεσε θύμα ανθρωποκτονίας και δεν υπήρξε κανένα είδου έρευνα του αγκλήματος, μόνο ατιμορρησία, οπότε αυτό απαιτούμε, απαιτούμε δικαιοσύνη και ήταν η γυναίκα μια φεμινίστα δημοσιογράφος. Υπέστη επιθέσεις, υπέστη απειλές, ακριβώς γιατί ζήτησε δικαιοσύνη και το θάνατο τη κόρη τη, Ε, κάτι άλλο, ένα άλλο φαινόμενο με τάση είναι η αύξηση της στρατιωτικοποίησης και η αύξηση των πολύ μεγάλων έργων για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Στο ΟΑΞΑΚ έχουμε πάρα πολύ αιωλική ενέργεια, ξυλία, μέταλλα και στο ΟΑΤΕΠΕΚ εκεί έχουμε αιωλικά πάρκα από την Ευρώπη και από άλλους και είχαμε εκεί τρεις ε, ακτιβιστές οι οποίοι δολοφονήθηκαν το 19. Στην περιοχή αυτή είναι επίσης είχαμε φαινόμενο στρατιωτικοποίησης που συνοδεύθηκε από ε, διχασμό στην ε, κοινωνία. Και όταν έρχεται ο στρατός στις πόλεις φοβούνται να βγουν οι γυναίκες και τα παιδιά γιατί έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις ε, ε, σεξουαλικής βίας όπως οι Φερνάντες και η Ροσέντο στην πολιτεία Γκερέρο. Ε, μια τρίτη τάση, ένα τρίτο φαινόμενο είναι η ατιμορρησία. Στις περισσότερες επιθέσεις οι ένοχοι δεν ε, συλλαμβάνονται παρά το ότι έχουν ε, εντοπιστεί. Και πολλές φορές η έρευνα που γίνεται ε, δεν λαμβάνεται υπόψη το ότι το θύμα ήταν ακτιβιστής. Το κονσόρτσιουμ αυτό της ΟΑΞΑΚΑ έχει υποστεί πάρα πολλές επιθέσεις και είχαμε επιθέσεις στα γραφεία, στα σπίτια ε, τα τελευταία 8 χρόνια και παρά το ότι έχουν γίνει δημόσιες ε, ε, καταγγελίες, αυτές όλες οι επιθέσεις δεν τιμωρήθηκαν. Επίσης είχαμε συκοφαντία στα μέσα ενημέρωσης και αμάυρωση της οργάνωσης μέσω του ίντερνετ. Οπότε το πρώτο θέμα είναι η ποινικοποίηση. Επίσης ε, όπως είπαν και οι συντρόφισσες από τις άλλες χώρες. Στο Μεξικό το, το 19 είχαμε α, πάρα πολλές αυθαίρετες συλλήψεις των ε, ακτιβιστών και ακτιβιστριών. Κυρίως άνδρες είναι αυτοί ε, που είναι ακτιβιστές, οπότε επιτίθενται στις γυναίκες τους, στις συντρόφισσες τους πολλές φορές έχουμε για τις ακτιβίστριες υποχρεωτικό εκτοπισμό και οι σύντροφοί τους ε, είναι μακριά από αυτές τις γυναίκες γιατί είναι σε κάποια μακρινή φυλακή. Η Ολάντα Κρούθ μια τέτοια περίπτωση ε, σε σχέση με έναν άλλον ακτιβιστή, σύντροφό που κρατήθηκε, ε, φυλακίστηκε επί 9 χρόνια και πριν από ένα μήνα σε είχε στείλει μια καταγγελία και οι βασικές επιθέσεις για αυτές τις ακτιβίστριε είναι ε, η δυσφήμιση, ολόκληρες ε, καταγγελίες δυσφήμισης, απειλές, επιθέσεις που είναι σεξιστικού χαρακτήρα και πολλές φορές ε, χρησιμοποιούν σεξουαλικά στοιχεία, κάνουν φωτομοντάζ, κάνουν στα κοινωνικά δίκτυα ε, τέτοιες τη δυσφήμισης ε, και χρησιμοποιούν την ηρωνία και κακόγουστα αστεία εις βάρος τους και όλα αυτά ε, γίνονται συνεχώς πάλι και πάλι στην ε, περιοχή αυτή που σας αναφέραμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, τώρα η τελευταία μας προσκεκλημένη είναι η Όλγα Αραούχο, εάν προφέρα σωστά το όνομά σας, προέρχεται από την Κολομβία. Καλησπέρα σε όλους, σε όλες, σε όλους τους ε, βουλευτές. Ονομάζομαι Όλγα Αράχο Κασανόβα και είμαι Κολομβιανή. Θα σας μιλήσω για μια περιοχή όπου η Νομαδέσκ, η οργάνωσή μας, ασχολείται με αυτό το κομμάτι της χώρας ε, στα νοτιοδυτικά, ρίνιο Κάουκα, Βάγε και Ουίλα. Αυτές είναι οι υποδιαιρές της ε, περιφέρειας αυτής. Στην ε, περιοχή αυτή έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες για την Κολομβία, διότι ο πληθυσμός εκεί αποτελείται από αυτόχθονες και από Αφροαμερικανούς στην πλειοψηφία τους. Και υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε αυτή την φάση για την περιοχή μας. Υπάρχει η οργάνωση στεγανή και υπάρχει και έντονη κινητοποίηση γιατί θέλουμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, να να αμυνθούμε ενάντια σε διάφορα φαινόμενα που συμβαίνουν. Αυτά γίνονται επομένως στο βορρά της περιοχής Κάουκα και στην Μποναβεντούρα. Εκεί υπάρχουν τα εξής σημαντικά χαρακτηριστικά. Η Κάουκα κατοικείται από αυτόχθονες πληθυσμούς και από κοινότητες νέγρων. στο πρώτο τμήμα της σήμερα. Υπάρχει κάτι που δεν δεν υπάρχει πουθενά άλλο, αλλά στην Κατατούμπα υπάρχουν τα ίδια και στην Βόρεια ε, Ακτή και στην Αμαζονία. Υπάρχουν υπάρχουν προβλήματα. Όμως, τέλος πάντων, εκεί στην Βόρεια Κάουκα τώρα, η κατάσταση που επικρατεί είναι, μια, είναι φαινόμενα δολοφονιών και διώξεων. σφαγές σφαγές του πληθυσμού και αυτό είναι επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Υπάρχουν παραστατιωτικές ε, ομάδες 98 με 2002 είχε ε, ενταθεί αυτό το φαινόμενο αλλά τώρα ξανά φούντωσε. Οπότε έχουν γίνει κάποιες ε, προσπάθειες ειρήνευσης ε, όταν είχαμε κάποιο είδους ε, εξεγέρσεις κατά του κράτους και τελικά κάναμε βήμα προόδου, μπορέσαμε να λύσουμε κάποια προβλήματα που είχαν να κάνουν με κοινωνικές ένοπλες συγκρούσεις. Όμως, όμως, όμως αυτό δεν πέτυχε 100% οπότε αυτό είναι αιτία πολλής δυσαρέσκειας, σε και χωριά. Είχαμε μια έκθεση του ΟΗΕ του περασμένου μηνό και μέχρι τον Οκτώβριο αναφέρεται αναφέρεται σε αυτή την έκθεση του ΟΗΕ για τον ΟΗΕ θεωρούμε ότι πρόκειται για ε, συμμάχους μας, αλλά είχαμε από αρχές της ε, χώρας 52 ανθρωποκτονίες και διάφορες παρασυλλογικές ε, ομάδες. Και αυτοί που σκοτώθηκαν ήταν άνθρωποι που αγωνιζόντουσαν για τον τόπο τους και τα δικαιώματά τους και είχαμε επίσης ε, τη δολοφονία 11 ηγετών τέτοιων κινημάτων. Τώρα οι γυναίκες σε αυτή την περιοχή. Οι γυναίκες στην περιοχή μας μπόρεσαν να συμμετάσχουν περισσότερο. Όσον αφορά την εκπροσώπηση στην κοινωνική οργάνωση. Όμως δεν υπάρχουν οι για να μπορούν να ασκήσουν τις αυτέ αυτές γίνεται. Είχαμε 19 αυτόχθονε που στη Βόρεια Κάουκα κατέβηκαν στις ε, εκλογές. Ε, σε δημοτικά συμβούλια, υποψήφιες ε, δύο, για δημαρχία, σε δύο, σε δύο πόλεις είχαμε τέσσερις υποψήφιες για το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κάουκα, αλλά δεν μπόρεσαν να ασκήσουν ε, τα δικαιώματά τους. Δεν γινόταν, δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε ε, ε, προεκλογική εκστρατεία. Οπότε, η Κριστίνα Μπατίστα είναι πιο πρόσφατα δολοφονημένοι. Αυτό μας προβληματίζει και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Πώς θα υπάρξουν εγγύησεις, πώς οι γυναίκες θα μπορέσουν να υπερασπιστούν τη ζωή τους και τη γη τους. να Βεντούρα. Άλλη περίπτωση. Εκεί χτυπάει η καρδιά της οικονομίας της χώρας. 65% της οικονομίας της Κολομβίας εδράζεται εκεί, σε αυτή την περιοχή. Επίσης είναι και πύλη προς την υπόλοιπη Νότια Αμερική. Έχουμε το πιο σημαντικό λιμάνι, αφορά πολλούς οικονομικούς κλάδους. Ε, επίσης ε, εκεί πέρα είναι πηγή ε, ποσίμου ύδατος που χρειάζεται για πάρα πολλούς. Πέντε φορέ έχουμε κάνει επίκουσε δράσει. Πέντε φορέ εκπέμψαμε το SOS και το Φεβρουάριο που είχαμε κάποια απόπειρα κατά κάποιων μαύρων γυναικών στη Βόρεια Κάουκα. Δύο στην Αμίγκα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας το κάνουν αυτό οι αυτόχθονε κοινότητε. Δύο φορέ κάναμε τέτοιε δράσει τον Ιούλιο, γιατί είχαμε κάποιε δολοφονίε, κάποιε απειλέ προ κάποιου ηγέτε και στη Βόρεια Κάουκα. Και επίση έγινε μια τέτοια πρωτοβουλία τον Αύγουστο, γιατί είχαμε πάλι κάποια απόπειρα ε, και δίωξη γυναικών που ασχολούνται με έναν φορέα για να μπορούμε να συμβιώσουμε με αξιοπρέπεια και ειρήνη. Οπότε για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν έχουμε τέτοιες πρωτοβουλίες που στέλνουμε δηλαδή το μήνυμα κινδύνου, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό η διεθνή κοινότητα να μπορεί ουσιαστικά κάτι να πει, να πάρει θέση, να μπορέσει να στηρίξει αυτές μας τις εκκλήσεις. Τέλος. Θα μπορούσαμε πολλά να σας πούμε, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι στις 12 Αυγούστου φέτος κάποιος ε, ηγέτης του κομματός μας, της φορέας μας τέλος πάντων, όχι, συγγνώμη. Κάποιος από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε στην Ποναβεντούρα. Ήρθε τόπου να δει ακριβώς υπό ποιες συνθήκες ζούμε στην Ποναβεντούρα. Στην Ίσλα Λαπάς, εκεί όπου έχουμε μία διεύρυνση, μία τέλος πάντων έργα ε, επέκτασης του λιμένος να δει τα προβλήματα με το νερό, να δει εκεί τι γίνεται όσον αφορά αυτή την επέκταση του λιμανιού της Μποναβεντούρα. Οπότε για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό όλες οι χώρες να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις γιατί θα πρέπει να υπάρξει καινούργια νομοθεσία γιατί α πούμε υπάρχει ένα νόμος που λέει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί, ότι θα πρέπει να γίνεται διαβούλευση για όλα τα έργα που γίνονται στον τόπο μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να λαμβάνεται υπόψη. Άλλο. Θα πρέπει κανείς να υποστηρίξει αυτές τις γυναίκες που δίνουν μάχη για την ζωή. Και αυτό θα πρέπει να το κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Ε, για τον ε, κόσμο που προέρχεται από τις χώρες που εμείς ε, προσωπούμε. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, λέει πρόεδρος, πάρα πολλές, αλλά θα δώσω τον λόγο στους συναδέλφους, στην Ιζαμπέλη Σλέρα από το ΕΛΚ. Καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μας είπατε, όσα μας περάψατε με ακρίβεια που αφορά την κατάσταση που είναι τόσο συγκλονιστική. Όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα παντού, θα πρέπει να στον προσοχή μας παντού όπου τα δικαιώματα καταπατούνται. Και το σούτο μάλλον καθώς έχουμε και τις γυναίκες σε πάρα πολλά μέρη που είναι οι πιο ευάλωτες. Και άκουσα τι είχατε να πείτε, άκουσα τι έχετε κάνει, τι δράσεις έχετε αναπτύξει και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά αυτά και πάλι ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε. Το πρόβλημα που μας περιγράψατε, όπως είπατε στην αρχή, είναι πρόβλημα όλων αυτών των χωρών και πολύ περισσότερων στην Λατινική Αμερική. Τι γίνεται, δεν μεταφράζονται αυτό που λέω. Συνεχίζω. Είναι θετικό που η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζονται και θα πρέπει να συνεργαστούν ακόμη περισσότερο. Έχω κάποιες ερωτήσεις για σας. Τι θέλετε να κάνει, ε, τι δράσεις διαλόγου θα πρέπει να κάνει το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή μας. Πώς θα μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. με τι ενέργειες θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε να σταματήσουν οι διακρίσεις. Έχετε βοήθεια εκεί, έχετε κάποιους που σας βοηθούν στη χώρα σας. Ε, βοηθά καθόλου το κράτος. Και είπατε και για την ατιμορρυσία. Τι μπορούμε να κάνουμε. Επίσης, μιλήσατε για πόλεμο σε επίπεδο επικοινωνίας, για παραπληροφόρηση, αν κατάλαβα καλά. Μπορούμε να αναπτύξουμε κάποιες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Και έτσι ούτως ώστε να έχει ακρίβεια η επικοινωνία. Και πάλι ευχαριστούμε. Σάντος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ε, καλύτερα να φορέσετε τα ακουστικά σας, λέει ο Μιλήτρη, θα μιλήσω, γιατί μιλώ πορτογαλικά. Θα ήθελα καταρχάς ε, να καλωσορίσω την ομάδα γυναικών αυτή που ήρθε με τόσο θάρρος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα για να προσπαθήσει να κινητοποιήσει την διεθνή κοινή γνώμη και την πολιτική βούληση των ε, πολιτικών ε, οργάνων. Και για να μπορέσουμε και εμείς να ενημερωθούμε για κάτι που συμβαίνει σήμερα στον κόσμο και που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία της γης ε, και το μέλλον της ανθρωπότητας διακυβεύονται. Θα ήθελα λοιπόν να αναγνωρίσω την τόλμη, το θάρρος των γυναικών αυτών στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν, ε, να προστατεύσουν τον τρόπο ζωής τους που με τη σειρά του προστατεύει και την ε, φύση, το περιβάλλον ε, και κατά συνέπεια και τη δική μας ζωή και την ανθρώπινη ζωή. Ακούσαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ε, όσοι υπερασπίζονται το περιβάλλον. Ακούσαμε τις απειλές που ε, ε, έχουν δεχθεί. Όταν δεν μιλάμε για γυναίκες, τα αντίπεινα είναι ακόμη πιο σκληρά. Το γνωρίζουμε αυτό. Γνωρίζουμε ότι ήδη οι γυναίκες είναι θύματα δίας και πάντα υποφέρουν περισσότερο σε καταστάσεις βίας. Ακόμη χειρότερη γίνεται η κατάσταση αν τολμήσουν να υψώσουν τη φωνή τους ε, και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ε, πιθανότατα να γνωρίζετε ότι οι πέντε ακτιβιστές δολοφονήθηκαν στην Κολομβία πριν λίγες μέρες, ε, μεταξύ των οποίων και γυναίκες. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο στην Κολομβία, συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Λατινικής ε, Αμερικής. Η αύξηση της βίας εις βάρος των ακτιβιστών είναι κάτι που αναγνωρίζεται σε όλες τις σχετικές εκθέσεις. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να στηρίξουμε τις ε, ΜΚΟ στις χώρες αυτές, ε, να ενδυναμώσουμε τις κοινότητες και τις γυναίκες αυτές, να τους δώσουμε λοιπόν τα μέσα να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τις κοινότητες ώστε να μπορέσουν να αντιστέκονται στις ε, πιέσεις που δέχονται. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μορφή βοήθειας που μπορούμε να παράσχουμε. Η Ιζαμπέλ όμως που πήρε το λόγο πριν ε, αναφέρθηκε στην ατιμορρησία. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω και για το θέμα αυτό. Δική μου εντύπωση είναι ότι στις κοινότητες αυτές ένα ε, αίσθημα ανυμποριάς ενισχύει την ιδέα ότι οι άνθρωποι που διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν διότι δεν ε, θα τιμωρηθούν ποτέ για αυτά που κάνουν. Είναι τεράστιο πρόβλημα για τις γυναίκες αυτές ακόμη και να έχουν πρόσβαση ε, στο δικαστικό σύστημα. Είναι πολύ δύσκολο να προσελκύσουν την προσοχή της αστυνομίας ή των αρχών στα προβλήματά τους. Θα, θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε τι προβλήματα αντιμετωπίσατε στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ε, τι προβλήματα αντιμετωπίσατε όταν προσπαθήσατε να απευθυνθείτε στο δικαστικό σύστημα και να ε, ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους, ε, τις ομιλητριές μας ε, και συμφωνώ με τους ότι είναι πολύ θαραλέο αυτό που κάνετε. Ε, δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω ότι βλέπουμε εδώ πέρα ένα μοτίβο σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ε, οι αυτόχθονοι λαοί γίνονται πολύ συγκεκριμένο στόχος και ιδιαίτερα οι γυναίκες ε, στις ε, ομάδες αυτές. Και αυτό άσχετα από τα ποια κυβέρνηση ε, υπάρχει. Το είδαμε αυτό όχι μόνο στις δικές σας χώρες, το είδαμε και στη Βραζιλία και, και τη Βενεζουέλα, όπου πρόσφατα συνομιλήσαμε με αυτόχθονες λαούς. Και μου φαίνεται ότι όχι μόνο ε, οι κυβερνήσει θένε, υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Έχουμε τη βιομηχανία εξόριξη ε, που αναζητεί πρώτες ύλες, ε, ιδιαίτερα χρυσό που συχνά βρίσκεται σε περιοχές αυτόχθονων κοινοτήτων. και όπου οι αυτόχθονες ε, κοινότητες ε, προσπαθούν να προστατεύσουν και το περιβάλλον από τέτοιες ε, δραστηριότητες. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που ανέφερε μια ομιλήτρια, που είναι ο ρόλος των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων εξόριξης εν μέρει από ευρωπαϊκές χώρες που ε, έχουν επιχειρήσεις ε, στις περιοχές σας ε, και που από τις κυβερνήσεις να διευκολύνουν τις δραστηριότητές τους. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να ασκήσουμε πίεση στις επιχειρήσεις αυτές. Εμένα με ενδιαφέρουν θέματα όπως είναι η ευθύνη της αλυσίδας ε, προμήθειας, κάτι που έχουμε συζητήσει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γενικά με ενδιαφέρει η ε, ε, επιχειρηματική ευθύνη, ώστε να γνωρίζουμε ότι τα προϊόντα που καταναλώνουμε εδώ στην Ευρώπη δεν είναι αιματοβαμμένα με το αίμα των αυτόχθονων κοινοτήτων. Ευχαριστώ πολύ, Χάιτι Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να εκφράσω ε, την εκτίμησή μου ε, στο όνομα της πολιτικής μου ομάδας ε, για τις ενέργειες σας στην περιοχή σας. Έχοντας ακούσει αυτά που είπατε, δεν, χρειάζεται, δεν χρειαζόμαστε άλλα επιχειρήματα για το γιατί χρειαζόμαστε, ε, γιατί χρειάζεται να εξετάσουμε ιδιαίτερα τη θέση των ε, γυναικών ε, ακτιβιστών. Ο Φινλανδός Υπουργός Εξωτερικών που είναι προεδρεύων στο Συμβούλιο οργάνωσε μια συνάντηση υπουργών στο Ελσίνκι τέλη Αυγούστου όπου προσκάλεσε γυναίκες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλοι συμφώνησαν ότι είναι απολύτως απαραίτητο για τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας ε, και ε, η κοινωνία των πολιτών να κάνουν ό,τι μπορούν για να υποστηρίξουμε το ρόλο των γυναικών υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είχαμε την Τερέζα Ριβέρα από το Ελσαλβαδόρ που είχε κρατηθεί και καταδικάστηκε λόγω αποβολής ε, και την καταδίκασαν ε, για φόνο. Αλλά αυτό πρέπει να το συζητήσουμε σε άλλο πλαίσιο. Απλά ήθελα να πω ότι αυτό που είπε μόλις η Ειρήνα είναι αυτό που θα πρέπει να εξετάσουμε ιδιαίτερα προσεκτικά. Την ε, δέουσα επιμέλεια των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ε, με δραστηριότητες εξόρυξης και γεωργίας. Θα παρακαλούσα να μου εξηγήσετε αν βλέπετε να υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και όσους λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις στη χώρα σας, διότι μερικές φορές το modus operandi, ο τρόπος που λειτουργούν είναι ότι οι τοπικές ελίτ ε, ευθυγραμμίζουν τη θέση τους με τις επιχειρήσεις, ενδεχομένως ε, για να δρέψουν και ιδιωτικό όφελος. Αυτό είναι ένα μοτίβο που βλέπουμε και συμφωνώ απολύτως με την Ειρήνα και πράγματι η Επιτροπή μας θα πρέπει να εξετάσει πώς μπορούν να λογοδοτούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταστροφή ε, του περιβάλλοντος όπου κατοικούν ε, αυτόχθονοι λαοί. Κάποιες ε, συγκεκριμένες υποθέσεις με απασχολούν. Έχουμε παρακολουθήσει με πολύ ενδιαφέρον την υπόθεση στην Ονδούρα της Ακοσάρκα, του φράγματος δηλαδή. Μετά από την ε, στιγμή δολοφονία της Μπέρτα Κασέρες. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τώρα τι γίνεται. Για μένα ήταν μάθημα το ότι και οι ε, οργανισμοί ανάπτυξης συχνά είναι συνένοχοι, διότι δεν μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματα των αυτοχθόνων. είδαμε Ολλανδικές και φιλανδικές επιχειρήσεις. Η δεύτερη με ερώτηση αφορά την ΟΑΧΑΚΑ. Ε, παρακολουθώ εδώ και χρόνια κάποια υπόθεση που... Ε, Ε, παρακολουθεί το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, την διπλή δολοφονία και έχω μεταβεί επανειλημμένα στην ΟΑΧΑΚΑ για να πάρουμε στοιχεία για την δολοφονία αυτών των δύο ακτιβιστών. Όπως όμως ακούσαμε είναι πολύ δύσκολο να αποδοθεί δικαιοσύνη στι υποθέσει αυτέ Αναρωτιέμαι ε, μήπως έχει ξεχαστεί η υπόθεση αυτή μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια στη Φιλανδία και στο Μεξικό. Σίγουρα θα έχουμε ε, ε, μια ε, τελετή μνήμης για την δολοφονία Φιλανδού και Μεξικανού υπηκόου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ροντρίγκες. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα-πρώτα να συμφωνήσω για τον σεβασμό, για την αναγνώριση της δράσης των προσκεκλημένων μας που ήρθαν στο Κοινοβούλιο για να μας εξηγήσουν με όσο γίνεται πιο ξεκάθαρο τρόπο όλες αυτές τις περιπτώσεις παρενόχλησης, ε, τις περιπτώσεις επίθεσης που ήρθαν και ως ακτιβίστες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και όπως εξήγησαν, ε, πρόκειται για πολύ συγκεκριμένε ενέργειε που αφορούν ακριβώς το ότι είναι γυναίκες και το ότι δίνουν αγώνες ε, ούτω ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι δικαιώματα που αφορούν τους ανθρώπους. Και ε, είχαμε κάποια, κάποιο θέμα όσον αφορά την προστασία για τους διάφορους τρόπους, για τους διάφορους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για να επιτεθούν στις ε, ακτιβίστριες. Ε. Ναι, οι γυναίκες είναι οι πρωτοπόροι του, του ακτιβισμού. Οι, οι γυναίκες, οι σύζυγοι, οι κόρες. Πεςτε μας δύο λόγια πάνω γι' αυτό. Τι γίνεται και τι γίνεται. Ε, οι άντρες σας υπερασπίζονται, οι σύζυγοι, οι γη σας, τα παιδιά σας σας στηρίζουν, σας βοηθούν, σας υποστηρίζουν. Επίσης, για πέστε μας, όσον αφορά τη δικαιοσύνη και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη με συγκεκριμένες επιθέσεις, ε, τι γίνεται, υπάρχουν συγκεκριμένα εμπόδια, φραγμοί για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη δηλαδή, ε, τι γίνεται όσον αφορά τις καταγγελίες για την παραβίαση των δικαιωμάτων. Επίσης, πώς βλέπετε το θέμα του ότι στα διεθνή πρωτόκολλα προστασία των ε, ακτιβιστών των δικαιωμάτων θα πρέπει ακόμα πιο ρητά να προβλέπεται η διάσταση του φύλου, ανισότητα, διακρίσεις, αποκλεισμοί. Επίσης, πέστε μας παρακαλώ δεν είναι πρώτη υποχρέωση ενό κράτου να υπερασπίζεται του πολίτε του. Θα πρέπει όμω και η διεθνή κοινότητα να τηρήσει αυτή την υποχρέωση. Οπότε θέλω να μου πείτε δύο λόγια για, την, για τις μεγαλύτερα, τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν ε, οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ στις χώρες σας. Τι σχέση έχετε με αυτούς τους φορές, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και να βοηθείτε περισσότερο. Βέβαια είναι και το θέμα της ειρήνευσης της Κολομβίας, είναι αυτή η συμφωνία που περιέχει πάρα πολλές ρήτρες για την ισότητα των φύλων. Πώς έχουν τα πράγματα, πώς ε, υλοποιείται αυτή η συμφωνία, η ειρήνευση. Δεν θέλω να λύτω λόγο. Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. για την τελευταία ομιλία. Έχουν αυξηθεί οι δολοφονίες κατά γυναικών, κατά των ακτιβιστριών και όσον αφορά τους αυτόχθονες. Είναι και αγωνίζονται τώρα περισσότερο, είναι περισσότερες ακτιβίστρες τώρα από ό,τι στο παρελθόν όσον αφορά τα θέματα του περιβάλλοντος. Υπάρχει περισσότερος κίνδυνος Ας πούμε βλέπουμε τι γίνεται με τα δίκτυα των ε, ε, ναρκωτικών στη χώρα σας, ε, γιατί εκεί οι θύτες είναι οι άντρες και θύματα οι γυναίκες. Πολλές φορές εσείς πλέον την ύφη γιατί είσαστε οι μητέρες ας πούμε, οι σύζυγοι αυτών που μπλέκουν με αυτά τα δίκτυα. Πέστε μας λοιπόν τι γίνεται που είσαστε ως γυναίκες οι στόχοι ε, και έτσι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος. Μας μίλησατε για τη διαβούλευση, τι γίνεται με τη διαβούλευση με τους αυτόχθανες για την εκμετάλλευση της γης τους και των πόρων τους. Δεν θα πρέπει να υπάρχει, όχι διαβούλευση, να υπάρχει σύμφωνη γνώμη. Γιατί η διαβούλευση πάνε να πει γνωμοδότηση και όχι απόφαση ε, για την αξιοποίηση της γης κάποιου κόσμου. Μήπως επιστώνεται ότι είναι ανεπαρκής η διαδικασία της διαβούλευσης. Έχετε το λόγο. Να αρχίσουμε με εσάς. Ευχαριστώ. Σε σχέση με λαοσά, ακούσαμε όσον αφορά ε, την ε, αντοχή μας. Ναι, βέβαια, θα πρέπει να βοηθηθούν οι γυναίκες ε, στις αυτόνομες κοινότητες. Ναι, γιατί είναι θέμα του Ιανουαρίου του 2018. όσον αφορά τις μοχέρες, την ισότητα των φίλων, τη δικαιοσύνη για το κλίμα. Το κείμενο αυτό του Κοινοβουλίου λέει ότι θα πρέπει κανείς να θωρακίζει τις γυναίκες και να φροντίζει και άλλα ζητήματα, πώς θα υπάρχει περισσότερη πρόσβαση όσον αφορά τη γη και θα πρέπει επίσης να υπάρξουν εγγυήσει όσον αφορά την λήψη αποφάσεων. Είναι ψήφισμα του Κοινοβουλίου και θα μπορούσε να μετατραπεί σε πρόταση, να δώσετε εσείς μια συνέχεια σε αυτό. Να δούμε τι γίνεται, πώς υλοποιείται, τι μέτρα λαμβάνονται συγκεκριμένα. Τώρα, όσον αφορά το πώς θα μπορούσε να πιέσει τις επιχειρήσεις στο Ισπανικό Κοινοβούλιο, όσον αφορά το πρόγραμμα δράσης για δικαιώματα και δημοκρατία της Ένωσης που είναι τώρα σε διαδικασία αναθεώρησης και διαβούλευσης κάτι θα μπορούσε να κάνει το Κοινοβούλιο είναι να εξετάσει εάν η Ένωση ενημερώνει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. εάν υπάρχει εποπτεία του αν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα τους επιχειρήσεις και σε σχέση με το δικαίωμα στην διαβούλευση. Ακριβώς, το κλειδί εδώ είναι η σύμφωνη γνώμη. Υπάρχει επίσης και το δικαίωμα στην αυτοδιαβούλευση, που είναι θέμα της αυτοδιάθεσης των λαών και αφορά και τους αυτόχθονες σε πολλές χώρες της ε, ε, Αμερικής και σε πολλές χώρες όπως το Μεξικό προβλέπεται ένα τέτοιο δικαίωμα αυτό διαβούλευσης. Οπότε λαμβάνεται υπόψη αυτό το δικαίωμα σε πολλές περιπτώσεις. Τώρα, όσον αφορά ε, τους Καρίνιο και Τζάκολα, σε αυτά τα εγκλήματα όντως υπήρχαν πάρα πολλοί στη δικαιοσύνη και ατιμορρησία. Και στο Μεξικό τα ξέρουμε τα θέματα γιατί η Καρίνιο ήταν ε, ιστορική, σημαντική ακτιβίστρια με μεγάλο ειδικό βάρος στην κοινωνία. Οπότε ε, έκανε πάταγο η δολοφονία της στην κοινωνία. Όμως μιλάμε για τρομερή ατιμορρησία. Έχουμε ένα σωρό επιθέσεις κατά ακτιβιστών που δεν τιμωρούνται. Άλλοι, κάποιοι τιμωρούνται, αλλά γενικά το μοτίβο είναι αυτό, η ατιμορρησία. Και όσον αφορά την ατιμορρησία, θέλουμε να παρέμβει σε αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση οι πρεσβείες, αντιπροσωπείες της Ένωσης έχουν μηχανισμό. Υπάρχει διαδικασία να έρχονται σε επαφή με τους ακτιβιστές και να υπάρξουν ε, βαθιές αλλαγές. Και οι δροματικές σας αποστολές να παρακολουθούν ε, από κοντά το τι γίνεται. Έχουμε ένα σωρό προτάσεις τώρα. Να γίνει κάποια ανάλυση από αμερόληπτους φορείς για αυτές τις ε, επιθέσεις. Τρίτες χώρες που κάνουν ε, τις σχετικές έρευνες να διερευνηθεί κατά πόσον λαμβάνουν υπόψη το ότι τα θύματα αυτών των εγκλημάτων είναι ή αυτόχθονες ή γυναίκες ή και τα δύο. Εσείς θέλετε να πείτε κάτι για τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. Έχω εδώ κάποιες απαντήσεις. Πρόσβαση στην ε, δικαιοσύνη, στην Ονδόρα. Λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Πολλές φορές το πρώτο που απαιτούν από εμά είναι το σώμα μας για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην ε, δικαιοσύνη. Το σώμα μας, ούτως ώστε να υπάρξει δικαιοσύνη. Επίσης, ρωτήθηκε κάτι άλλο. Αν μας βοηθάει κανένας. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες προστασίας. Και πολλές φορές όμως αυτός ο μηχανισμός αποσκοπεί στο να ζητήσει πληροφορίες για τη δραστηριότητά μας, αντί να μας βοηθάει. Οπότε μας, μας έρχεται πανικός φόβος όταν έρχονται αυτοί δίθεν να βοηθήσουν και πρέπει να τους αναπτύξουμε το θέμα μας. Ε, αντί να βοηθήσουν μέχρι και μας σκοτώνουν αυτοί που ε, αποτελούν κομμάτι του μηχανισμού βοήθειας. Σε ένα χωριό έγινε αυτό, είχαμε δύο δολοφονίες με, αυτό την, ε, με αυτόν τον τρόπο. Αντί να βοηθηθεί δηλαδή αυτός ο κόσμος, υπέστη αυτό. Επίσης, όσον αφορά και τις ε, εταιρείε εξόριξης. Τι μπορεί να κάνετε. Θα πρέπει να χτυπήσετε το καμπανάκι, να καταλάβουν οι εταιρείε ότι γίνεται στη χώρα. να λάβουν υπόψη τι γίνεται σε πόλεις και χωριά. Μην νομίζουν ότι όλα είναι στρογγυλά για τελικά εμείς να υφιστάμεθα τα, τα πάντα από, από αρρώστιες. Να καταλάβουν, να καταλάβουν αυτοί τι γίνεται με τα έργα τους αυτά τα οποία ε, ότι θα πρέπει αυτά τα έργα να ωφελούν και τις κοινότητες. Γιατί στι περισσότερε περιπτώσει έχουμε καταστρέψει του περιβάλλον, έχουν καταστραφεί, έχουν ε, βρωμίσει τα, τα ποτάμια μα. Δεν το λαμβάνουν υπόψη. Τόσο νερό είχαμε, αλλά τώρα δεν έχουμε τίποτα. Μα πήραν και την άμμο. Πάντα ποτάμια. Έχουν μολύνει όλη τη χώρα. και τι υφίστανται επίση ε, ανήλικοι γυναίκε, ένα σωρό αρρώστιε ακριβώ από τέτοια, έργα και τα υδρο, υδροηλεκτρικά φέρει Αυτή η πώ το λένε τέλο πάντων. Και σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει ε, τομέα υγεία, δεν υπάρχει πολιτική υγεία. Οπότε στην Ονδούρα ούτε, ούτε υπάρχει κρατική πολιτική υγείας και το αντίθετο, μας παίρνουν την υγεία μας. Οπότε, για την οικογένεια λίγα πράγματα γίνονται. Όταν υπάρχει όταν υπάρχει κάποιος ακτιβιστής, κάποια ακτιβίστρια, διαλύεται η οικογένεια, θα πρέπει κανείς να, φύγει από τη χώρα. Θα πρέπει να, δραπετεύσει από την ίδια του τη χώρα. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ναι. Ε, Όσον αφορά για την ατιμορρησία και την ερώτηση που κάνατε, στη Γουατεμάλα έχουμε κατά επανάληψη κάνει καταγγελίες, αλλά δεν έγινε τίποτα. δίνουμε όλα μας τα λεφτά σε δικηγόρους και λοιπά, αλλά... Αλλά... Μας φυλακίζουν. Αποφυλακιζόμαστε και μετά μας ξαναβάζουν τη φυλακή γιατί υπερασπιστήκαμε το δάσος, για παράδειγμα. Ή όταν ας πούμε αναπτύσσουμε δράση για τις εξωτερικές δραστηριότητε, για το ποτάμι. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα μας. ατιμορρησία, παρά τις καταγγελίες. Αναλωνόμαστε οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος. Τι μπορείτε εσείς να κάνετε, ρωτήσατε. Τι πρέπει κάτι να γίνει για τις επιχειρήσεις στη χώρα μας. Θέλουμε οι αντιπροσωπείες σας στις χώρες μας να κάτσουν και να καταγράψουν τι γίνεται σε χώρες, σε πόλεις και χωριά, τι γίνεται με τα ποτάμια. Δεν μας αφήνουν να πάμε στα ποτάμια μας, ούτε να ψαρέψουμε. δρολητικά έργα, οι καλλιέργειες ε, του αφρικανικού φίνικα. Άρα, να κάτσουν και να ελέγξουν τι γίνεται, να παρακολουθήσουν, να υποπτεύσουν. Γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά μας ως λαού. Υπάρχουν ιστορικά δικαιώματα, δικά μας επί της γης. Αλλά τίποτα δεν γίνεται. Να γίνουν σεβαστά αυτά τα ιστορικά δικαιώματα των λαών. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα η τελευταία είναι η Όλγα Αραούχο. Αυτό που χρειάζεται είναι το εξή. Τα είπαν και ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια παρακολούθηση των εξελίξεων και ακριβώ όπω είπατε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, τι συνέχεια δίνεται, αν θέλουν κάποιες λύσεις τι γίνεται στην ε, πράξη, τι γίνεται με την συμμετοχή των ε, κοινοτήτων και των γυναικών. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι καλά έχουμε αυτά τα ψηφίσματα, αλλά, αλλά αυτά μένουν στο χαρτί, δεν φτάνουν στις ακτιβίστες, δεν φτάνουν εκεί επιτόπου στον κόσμο. Και το ίδιο ισχύει και με το τι θα γίνει με το πρόγραμμα δράσης των δικαιωμάτων ε, από πλευράς των ε, κρατών μελών. Γίνει κάποιες διαβουλεύσεις, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτά πολλές φορές ε, καταστρατηγούνται. Έχουμε όσο με κάποιες εταιρείε εξόριξης που μιλάνε για προ, προ, προηγούμενη σύμφωνη γνώμη αλλά τι πάνε να πει αυτό, να πάμε να βρουν κάποιον οποιονδήποτε και κάποιο οποιοδήποτε λέει ναι εντάξει έχετε το πράσινο φω. Όχι, χρειάζεται μια ελεύθερη διαδικασία διαβούλευση. Οπότε υπάρχουν ε, αυτέ οι διαδικασίε που σημαίνουν εποπτεία, σημαίνουν διαβούλευση, διάλογο και όλα αυτά θα πρέπει να ελοποιούνται πολλέ φορέ τι υποσχέσει δεν τι κρατάει η κυβέρνηση. Αυτό θα πρέπει να δούμε. Τι γίνεται, αν τηρείται στις χώρες που συζητούμε, στις χώρες μας η νομοθεσία. Και από πλευρά κοινοβουλίου θα πρέπει αυτό να λυθεί Τι γίνεται με την νομοθεσία. Και να υπάρχει στην ουσία διαβούλευση και επικοινωνία με τις γυναίκες, με τις κοινότητες, με αυτούς που πραγματικά θίγονται και εμπλέκονται. Γιατί πάρα πολλά ε, γίνονται και μένουν εδώ, στα δεσμικά όργανα. Και να δώσουμε τον λόγο στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Merci beaucoup. Ε, je vais pas. Ε, ε, I will not take lots of time. I would. Christo, δεν θα μακρηγορήσω. Απλώς θέλω να πω ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται ένα νέο επεξηγηματικό σημείωμα το οποίο θα κατευθύνει τις δράσεις μας και θα αφορά ιδίως τις ακτιβίστρες υπερασπίστρες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο πλαίσιο αυτό στις 3-4 Δεκεμβρίου εδώ στις Βρυξέλλες διοργανώνουμε το Ευρωπαϊκό ε, Φόρουμ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δίκτυο ε, οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τίτλο και αντικείμενο την προστασία των ακτιβιστών ε, του περιβάλλοντος ε, και με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Πάντως σας ξαναευχαριστώ θερμότατα που ήρθατε εδώ. Θα κάνουμε ένα μια δοκιμή για να δούμε αν λειτουργεί καλά η σύνδεσή μας με την Συρία. Θα δούμε αν μπορούμε να συνδεθούμε. Bonjour, vous nous entendez bien Bonjour. Vous m'entendez On vous entend, on vous voit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 να το Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με το πέμπτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Αποκινούμε την Επιτροπή Ανάπτυξη, ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρωπιστική κατάσταση στη βορειοανατολική Συρία. Έχουμε μια σύνδεση μέσω Skype με δημοσιογράφο. Η σύνδεση είναι καλή, όπως διαπιστώσαμε, οπότε θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Υπό το φως και των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Τουρκίας, που ξεκίνησαν έπειτα από την ακατανόητη απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή, και θέλουμε βεβαίω ε, να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρωπιστική κατάσταση έτσι όπω έχει διαμορφωθεί. Θέλω να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, ο οποίος θα συμπροευρεύσει την, τη συνεδρίαση μαζί με εμένα. και του δίνω και το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Αρένα. Σας ευχαριστώ που διοργανώνετε αυτή την ε, ανταλλαγή απόψεων και που γίνεται από κοινού με τη δική μας Επιτροπή. Ο πρόεδρος μας, ο κ. Στομπέ, δυστυχώς ε, δεν μπόρεσε να έρθει, διότι υπάρχει ταυτόχρονη ε, συνεδρίαση των Επιτροπών ΤΕΒΕ και ΑΦΕΤ με τον Πρωθυπουργό του Σουδάν, οπότε είναι τιμή μου που εκπροσωπώ εγώ τον κύριο Τομπέ ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Υπογραμμίζω και εγώ αυτό που είπε η κυρία Αρένα ε, σχετικά με την ακατανόητη απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων και την ε, ε, μετέπειτα στρατιωτική εισβολή των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων που καταδικάστηκε και από το ψήφισμα στην Ολομέλεια πολιτικές ανησυχίες ε, και ανθρωπιστικές ανησυχίες ε, που προκάλεσε η στατική αυτή επιχείρηση είναι πολύ σημαντικό θέμα, γι' αυτό και θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Θέλω να ε, επικεντρωθώ στις ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές διαστάσεις αυτής της εισβολής. 250.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν λόγω της εισβολής αυτής. Ένα μήνα μετά, 100.000 άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι στην, ε, σε διάφορες περιοχές της Συρίας, το ε, ε, Χαλέπι, την Ράκα, καταστράφηκαν σχολεία, νοσοκομεία, οι άνθρωποι ζουν σε εξαιρετικά επισφαλείς συνθήκες. Είναι τεράστιο το πρόβλημα εν ώψη και του επερχόμενου χειμώνα που μπορεί να είναι πολύ σκληρός στην περιοχή. Ε, γι' αυτό και έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία ε, παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, τροφίμων και ρουχισμού στους ανθρώπους. Δεύτερον, Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα μη κυβερνητικέ οργανώσει και υπηρεσίε του ΟΗΕ στην ε, βορειοανατολική Συρία, η στρατηγική αυτή εισβολή είχε μεγάλες επιπτώσεις, καθώς πολλοί διεθνείς εργαζόμενοι έχουν εγκαταλείψει, των μη κυβερνητικών οργανώσεων έχουν εγκαταλείψει την περιοχή. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί ασφαλείας ε, που έχουν εμποδίσει την παροχή ανθρωπιστικής και αμυντικής βοήθειας. Μόλις χθες ένας εργαζόμενος μη κυβερνητικής οργάνωσης τραυματίστηκε σοβαρότατα έπειτα από επίθεση που ε, υπήρξε εναντίον του οχήματος που τον μετέφερε. χρειάστηκε να παρέμβουν ε, δυνάμεις για να ε, παράσχουν αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει γρήγορα να αρθούν όλα τα εμπόδια ώστε να παρασχεθεί η βοήθεια σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο. Και τώρα θέλω να ακούσουμε από τους ε, προσκεκλημένους μας πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί επί τόπου. Σας ευχαριστώ. Όπως είπα πριν, από τότε που έγινε η τουρκική εισβολή και επιστροφή στην περιοχή των, του Συριακού στρατού έφυγαν οι οργανώσεις και έχουμε πάνω από 4.000 σε κατάσταση πηγούς ανάγκης. Και για αυτό και ε, εξετάζουμε το θέμα πλευράς δικαιωμάτων και ανθρωπιστικής πλευράς. Οπότε, θα δώσουμε ευθύ αμέσω τον ε, λόγο στο Ραφέλ Λεμπιουρζά. Βρίσκεται στην Συρία και πρόκειται να μας καταθέσει την μαρτυρία του για αυτά τα οποία ζει επί τόπου. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον και μετά να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Ραφαέλ, έχεις το λόγο. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Σας πω πώς έχουν τα πράγματα. Ευχαριστούμε και τους διοργανωτές που μας προσκάλεσαν και τους ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα που κατέστησαν εφικτή αυτή την επικοινωνία. Έτσι, νομίζω θα φωτίσουμε το πρόβλημα. Μιλούμε για τον κουρδικό πληθυσμό που βρίσκεται εδώ, τις αρχές που είναι πλάκησαν εδώ, που ήταν στην πρώτη γραμμή του πολέμου κατά του Ισλαμικού κράτους. Έγινε αυτή η ακατανόητη απόσυρση των Αμερικανών και όλα αυτά λίγες μέρες τα βρήκανε με τους Αμερικανούς οι Τούρκοι λίγες μέρες πριν εισβάλλουν. Τώρα εδώ ο κόσμος είναι αγανακτισμένος κατά του ΝΑΤΟ, κατά της δύση. Τους θεωρούν συνένοχους αυτά που γίνανε, που διαλύθηκε όλη τους η άμυνα. Και η τρώνε υπεράσπιση εναντί των Τούρκων που τους αγκατέλειψαν οι Αμερικανοί. Και κάθε μέρα εδώ και ένα μήνα ζω τις εξελίξει εδώ. Πρώτα πρώτα είχαμε σε όλο το μήκος των συνόρων συγκρούσεις παντού σε όλες τις παραμεθόριες πόλεις είχαμε συγκρούσεις. Είχαμε εκτοπίσεις, αναχωρήσεις μαζικές. Μερικοί ξανά ήρθανε. Γενικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί ακριβώ όπως λέχθη στην αρχή από την Πρόεδρο, σήμερα δεν υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια προς εδώ, όπως θα όφελουν να υπάρξει. Έχουν φύγει η ΜΚΟ. Όλο. Πρόσφυγες. Αυτά είδα. Πρόβλημα διατροφής των παιδιών. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση για αυτά τα παιδιά σήμερα. Δύσκολη η επιβίωση. Πρόβλημα διατροφής, πρόβλημα ε, από αρρώστιες που εξαπλώνονται και έχουμε πάρα πολλούς πρόσφυγες που έτσι κι αλλιώς υπήρχαν και πριν από αυτή την επίθεση, αλλά τώρα αυτοί βρέθηκαν ακόμα πιο στριμωγμένοι. Επίσης, κάτι άλλο πολύ εντυπωσιακό, ότι εδώ έχουμε τους Τούρκους, τους συνεργάτες τους, έχουμε κάποιους Ισλαμιστές που άλλαξαν στρατόπεδο ε, και έχει γίνει τρομερή καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ. Με τα μάτια μου είδα βομβαρδισμούς χωρίς διακρίσεις. Ήμουν στο Τελτάμερ, εκεί που κατοικούν Κούρδοι, Χριστιανοί και Χριστιανοί και εκεί έγιναν αυτοί οι βομβαρδισμοί και ήμουν με έναν συνάδελφο δημοσιογράφο και έριξαν βόμβα 30 μέτρα από εκεί που βρισκόμασταν. Χωρίς να υπάρχουν εκεί και τίποτε μαχητές. Δεν υπήρχε στρατιωτικό στόχος εκεί. Πρόκειται για τρομοκρατία δια του βομβαρδισμού. Στην αρχή των συγκρούσεων, είχαμε αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χτυπήθηκαν πάρα πολλοί άοπλοι. Πάνω από 250 ήταν οι πολίτες οι οποίοι σκοτώθηκαν από την αρχή της ε, τουρκικής επίθεσης. Οπότε μέσα σε αυτό το σκηνικό έχουμε πολλούς τραυματίες, πάνω από 2.000 και 200 με 250 χιλιάδες που απειλούνται. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Είχαμε και βομβαρδισμούς ε, σε χώρους που υπάρχει πόσιμο νερό. Και μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδων που έχουν πρόβλημα παροχής ύδατος. Δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Έχουμε ένα σωρό στρατοφυλακές ε, τζιχαντιστών που λαιλατούν, ε, εκκλησίες. Ε, συγγνώμη που δεν σας τα λέω τόσο τακτικά, αλλά σας τα λέω εκ των ενόντων. Και επίσης υπάρχει και θέμα εθνοκάθαρσης, σημαντικό ο Ερντογάν πρόσφατα είπε ότι δεν έχουν θέση εκεί οι Κούρδοι. Οι Άραβες ε, έχουν θέση εκεί, είπε, μια που έχουν συνηθίσει την έρημο. Πρόκειται δηλαδή για εθνοκάθαρση εκ Γι' αυτό ότι ασκούν τρομοκρατία οι Τούρκοι και οι ουρές τους. Χτυπήσαμε δύο σημαντικές πόλεις. Ε, λένε ρεζερβέ και έτσι σημαδεύουν κάποιες ε, κατοικίες και έτσι απαλωτριώνουν, ε, κατάσχουν κάποια σπίτια, σπίτια χριστιανών, αυτοί οι στρατοφυλακές. Και μιλάω τώρα ότι χτυπιέται ο κόσμος που ήταν οι σύμμαχοί μας κατά του Ισλαμικού κράτους. Επίσης, έγιναν ε, απαγωγές. Ε, πιάσανε και με συνοπτικές διαδικασίες εκτέλεσαν κάποιους ε, νοσοκόμους του Ερυθρού Στρατού, συγγνώμη, του Ερυθρού Σταυρού. Και Επίση απάγουν κάποιους, ζητούν λίτρα της οικογένειάς τους, ε, ανακρίνουν τον κόσμο. Τέσσερι ε, Κούρδοι δημοσιογράφοι επίσης εκτελέστηκαν, όπως λέγαμε, βομβαρδίζουν ένα σωρό πόλεις, αστικές περιοχέ. Πολίτες. Καμισόντ, Κομπάνι, Τελαμπιά και, και σε άλλα μέρη. και στοχεύουν οι βόμβες τους χριστιανούς και Κούρδους, τους τρομοκρατούν. Επίσης υπάρχει η υποψία χρήσης χημικών όπλων στο Μενσουράν. Είχαμε κάποιον Σουηδό γιατρό, ο οποίος είναι ειδικό στα χημικά ξέρει για τα θέματα των δικαιωμάτων και είπε ότι αφού εξήτασε διάφορα θύματα, είπε ότι έχουν χτυπηθεί με χημικά. Και συμφωνούν μαζί του και διάφορες ανθρωπιστικές ε, οργανώσεις. Επίσης, έχουμε αυτέ τι παραβιάσει ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία και άλλο για το διεθνού δικαίου το έκανε η Τουρκία. Δεν σέβονται την ε, εκεχηρία που είχε συμφωνηθεί. Κάθε μέρα έχουμε ε, ακριβώ συγκρούσει. Χτυπιούνται στι ε, κουρδικέ πόλει πολίτε. Αλλά δεν φτάνουν μόνο αυτά. Η, η εισβολή οδήγησε σε αύξηση των επιθέσεων του Ισλαμικού κράτους. Σήμερα σκοτώθηκε ένας ιερέας Αρμένιος από το Ισλαμικό κράτος. Είχαμε 48% αύξηση των επιθέσεων του Ισλαμικού κράτους. Σημαντική αύξηση. Τις 10 δε πρώτες μέρες του Νοεμβρίου πάνω από 30 επιθέσεις. 300% σε σχέση με τις 10 πρώτες μέρες του Οκτωβρίου. Άρα, πολλαπλασιασμός των επιθέσεων του ΝΤΕΣ που είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Σήμερα είχαμε βομβιστικές επιθέσεις. Όλα αυτά από την τουρκική εισβολή. εθνική κάθαρση αυτό, εθνοκάθαρση εκεί που είναι οι Κούρδοι και οι Χριστιανοί. Επίσης συνάντησα ένα παιδί, ένα, ένα μικρό σύρο ε, που έχει τα, πάθει ψυχικό τραύμα από τους βομβαρδισμούς ε, έχουμε επίσης ε, από μεγάφωνα προσευχές κάθε φορά που ακάει το Αλάχου Άγμπαρ τρομοκρατείται. Άρα πρόκειται για βιομηχανία φόβου. Όλοι εκεί είναι σοκαρισμένοι από αυτήν την κατάσταση. Καταστροφή. Είπαμε επιθέσεις με στόχο την εθνοκάθαρση. Είναι σαφές. Όλα αυτά από τότε που άρχισε η επέμβαση. Επίσης, έχουμε και δολοφονίες πολιτών. Εγώ διαφόρων ηθινόντων, την Ευρύν Χαράφ, που ήταν ε, πρόεδρος ε, κάποιου οργάνου γουρδικού και στον ε, αυτοκίνητο M4 τη σκότωσαν οι Τούρκοι ενώ είχε μετακινηθεί ε, στα πλαίσια των καθηκόντων της και οι δολοφόνοι τράβηξαν βίντεο. Στην Τουρκία μιλούν για το ότι η αποστολή επέτυχε. οι τουρκικές αρχές ξέρουν απολύτως του τι γίνεται, το τι κάνουν οι συνεργάτες τους. Σφαγές κατά του πληθυσμού. Εξαπλώνεται παντού ο τρόμος. εκτοπίζουν κόσμο και φέρνουν οικογένειες να τους άλλες να αντικαταστήσουν αυτούς που εκτοπίζονται. αμερικανικά και ευρωπαϊκά όπλα χρησιμοποιούν. Κυκλοφορούν και φωτογραφίες από τον στρατό του Ισλάμ που είναι μία από τις στρατοφυλακές που πολεμούν με τους Τούρκους. Είχαν ένα Λέοπαρντ γερμανικό, ένα τάγκ Λέοπαρντ και το χρησιμοποιούσαν σε επιχείρηση κατά των Κούρδων. στο Χαλέπι, βάζουν ε, χμάλο τους ε, σε κλουβιά και τους πάνε γύρω γύρω για να τους ταπεινώσουν. Ε, αυτές οι πρακτικές του φόβου. Τα ίδια κάνουν οι τζιγαντιστές που χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά, είπαμε και αμερικανικά όπλα για τα εγκλήματά τους. Και όπως είπαμε στην αρχή, είχε υπάρξει υπόσχεση της διεθνούς κοινότητας για προστασία των Κούρδων. Βέβαια σήμερα ε, έλαβε μέτρα η διεθνής κοινότητα σε σχέση με την πώληση των όπλων. Και ο κόσμος όμως εδώ πιστεύει ότι η Ευρώπη λέει πολλά αλλά δεν κάνει τίποτα. Οπότε, Είπαμε, πρόκειται για εθνοκάθαρση ε, και έχουν φύγει πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Δεν υπάρχει έλεγχος και ο κόσμος φοβάται, δεν εμπιστεύεται τις αρχές. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται από μεγάλη ένταση, είμαστε μεταξύ σφύρας και άκμονας και ε, θεωρούν ε, ότι δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις. Από ανθρωπιστικής πλευράς και ανθρωπίνων δικαιωμάτων η κατάσταση είναι καταστροφική. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις. Ε, Πρόεδρος, ευχαριστούμε να δώσουμε το λόγο στους άλλους ε, δύο που θα μιλήσουν. Αν μπορείτε μείνετε στο ακουστικό σας και να ακούσετε μετά τι θα πούν τα μέλη της Επιτροπής μας. Συμφωνείτε? Συμφωνεί, λέει ο Ραφαήλ. Λοιπόν, δίνω το λόγο στον Μιάκ Πιερινή για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια συνολική εικόνα και μετά στον ε, Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ακούσαμε από την πρώτη γραμμή. Εγώ ε, θα σας μιλήσω ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμος σήμερα, πρώην πρέσβης στην Τουρκία και στη Συρία. Γιατί έγινε αυτή η στρατιωτική εισβολή από την πλευρά της Τουρκίας και τι περιμένουμε στο μέλλον. Πρόκειται για λογικό απότοκο των όσων είχαν προηγηθεί ε, το 2016 και 2018 όταν έγιναν δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας, οι οποίες είχαν ως στόχο να ε, προλάβουν την ε, μετακίνηση συριακών ε, στρατιωτικών μονάδων προς τα δυτικά. Και η συγκεκριμένη προσπάθησε να αποκόψει το κομπάνε από την Τζαζίρα. Αυτή ήταν η κατάσταση προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στην Συρία. Η τουρκική λοιπόν αντίληψη ε, εντάσσεται σε, αυτήν την, σε αυτόν τον ε, φόβο τον οποίος είναι ε, για τους Ροζάβα και τη Συρία που είναι κοινό φόβος σε όλα τα πολιτικά κόμματα και σε όλους τους πολιτικούς στην Τουρκία. Σε σύγκριση λοιπόν με τα όσα ισχυρίζεται η τουρκική ηγεσία δεν ε, ε, ελέγχει 440 χιλιόμετρα συνόρων. Μόλις 120 είναι τα χιλιόμετρα που ε, ελέγχει η Τουρκία γιατί επενέβησαν γρήγορα οι ρωσικές δυνάμεις. Η κατάσταση είναι ασταθής και καθόλου τόσο σταθερή όσο ήθελε αρχικώς η, η Άγκυρα. Πριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της Τουρκίας θα παραμείνουν στη Συρία έως ότου ε, αποσυρθούν όλα τα ξένα στρατεύματα συμπεριλαμβανομένων των ρωσικών. Και αυτό θέτει ένα νέο ερώτημα. Πρόκειται για προσωρινή στρατιωτική επιχείρηση ή πρόκειται για μόνιμη κατοχή. Τρίτον, πριν από... από τον Υπουργό Εσωτερικών και από τον Πρόεδρο ότι θα αρχίσει να στέλνει στην Ευρώπη τους τζιχαντιστές εκείνους που ήταν στην Συρία μέσω του, της επικρατείας θα τους στείλει στην Ευρώπη, το είπε σήμερα το πρωί ότι αυτό θα κάνει αυτή την εβδομάδα έτσι θα συνεχιστεί και όπως πολλοί γνωρίζουν έχουμε ήδη έναν τζιχαντιστή Αμερικανό ο οποίος απελάθηκε και αυτά έναν Δανό και έναν Γερμανό ε, μετά ε, από άλλου Γάλλου, Γάλλους, δηλαδή, έχουμε δηλαδή συνολικά 1200. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση στην οποία τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει, να βρίσκεται ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, Πολλέ χώρε μέλη τουλάχιστον πρώτα για μια στρατηγική ανοιχτή αντιπαράθεση με την Δύση, με την Ευρώπη. Και έτσι είχε γίνει ε, με τη Γαλλία όταν είχαμε κάποιο επεισόδιο, τυχαίο ή επίτηδες, το οποίο κατέληξε σε μια πολύ πιο ισχυρή αστυνομική επιχείρηση Γαλλίας ε, Τουρκίας, αλλά τώρα επίτηδες θέλουν να στείλουν τζιχαντιστές Ευρωπαίους. Και εκείνους δηλαδή που τους είχε αφαιρεθεί η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο πρόβλημα της Τουρκίας. Είναι θέμα διεθνούς δικαίου. Μα πώς γίνεται ένα κράτος να κάνει απάτριδα κάποιον υπηκό του. Επίσης, για πολλούς μήνες, η Τουρκία στέλνει στο βόρειο-ανατολικό τρίγωνο στην Συρία ε, από ένα μέχρι τρία εκατομμύρια από τους πρόσφυγες που βρίσκονται στο εδαφός της η Τουρκία. Αυτό Βέβαια είναι ανήκουστο, η, αλλά είναι, είναι αδύνατον σε αυτό το μικρό χώρο που κατέχει η Τουρκία. Άρα θα πρέπει τώρα να ψάξουμε να δούμε μήπως αυτό έχει ελαττήρια εσωτερικής πολιτικής. Τη, γιατί ε, θεωρεί η ηγεσία της χώρας ότι η αποτυχία στις δημοτικές εκλογές και στις πανελληνικές της Κωνσταντινούπολης ότι αυτό οφείλεται στην παρουσία των προσφύγων που θύμωσαν τον πληθυσμό. Φυσικά και ξέρουμε ότι αυτό δεν έχει σχέση. Οφείλεται στην κακή οικονομική κατάσταση της χώρας, οφείλεται ε, στην πτώση του κυβερνώντος κόμματος. Οπότε μέσα σε αυτή τη λογική θα πρέπει να γυρίσουν, λέει, όσο γίνεται περισσότεροι, να φύγουν πιο πολύ από τη χώρα, λέει η λογική της Άγκυρας. Ε, αυτά τα έχουμε απορρίψει και στο Συμβούλιο και εδώ το Κοινοβούλιο, αλλά εδώ πέρα αναδύονται πάρα πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν το ποιο θα πάει πού, από ποια, από ποια, από τι, τι, θα είναι αυτοί που θα πάνε και πού. Ε, να δούμε επομένω τι θα πει το Συριακό καθεστώς, ε, τι γίνεται, γιατί να τιμωρούνται ε, αυτοί που ήδη επέστρεψαν εκεί, κάποιοι φυλακίζονται, σε κάποιους έχουν πάρει τα σπίτια, τι θα γίνει με τις διεθνείς ε, συνθήκες, τι θα γίνει μια πολιτική συμφωνία, πώς θα υπάρξουν εγγύσει για την ασφάλεια αυτών που θα επιστρέψουν και πώς όλα αυτά με ποιο μηχανισμό θα ελεγχθούν. Πολύ σημαντικά θέματα. Γίνεται βέβαια ένα παζάρι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά θα πάνε σε κάποιες ε, συνομιλίες ε, μεταξύ Ερντογάν ε, και κάποιων ηγετών μέσα σε λίγες εβδομάδες στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Οπότε θα μας πει ότι αν δεν χρηματοδοτήσετε αυτή την επιστροφή, δηλαδή ε, το να φτιαχτούν κάποια κτίρια και δομές υποδοχής τέλος πάντων, τότε θα ανοίξουμε την πόρτα της εξόδου. Βέβαια, το θα ανοίξουμε την πόρτα σημαίνει κάτι πολύ περίπλοκο, μια περίπλοκη πολιτική ε, και η μεταφορά Αφγανών, Αιθιώπων, από την Ερυθρία τέλο πάντων, ε, προσφύγων όλοι αυτοί, από τις μαφίες που τώρα κυριαρχούν εκεί θα πάνε στην Ευρώπη. Φυσικά και αυτό είναι εκβιασμός. Αυτό είναι ένα παζάρι, είναι η διπλωματία του παζαριού. Αν θέλετε ακριβώς, ε, ε, ακριβώς όπως έγινε το 15-16 με τους πρόσφυγες. Αυτά τώρα ξανακάνουν. Αλλά ε, τώρα η βάση αυτού του παζαριού, αυτής της υπόθεσης, είναι αυτοί οι Ευρωπαίοι μαχητές. Bonsoir et merci pour nous donner, de nous accorder cette chance pour parler aujourd'hui et exprimer notre point de, vue, de, vue, de vue à vous. Μπορείτε να κάνετε αυτό, παιδιά. Το, το έχουν όλοι. Από τα γαλλικά. Τα παίρνουν τα γαλλικά. Όλοι. Δεν κάνουν όλοι. Τώρα δεν ακούγεται τίποτα. Όταν μόλις εγγύσεις πάρει σοκολάτα πάνω σου χρειάζεται. التي تكلم بها مخلصنا الرب وهي ذات اللغة التي نتكلمها اليوم نحن كسريان في مجتمعنا في سوريا. Le peuple syriaque araméen est l'un des premiers peuples à avoir cru en Jésus-Christ, l'un des premiers à avoir adopté ses idées et sa Ο αραμαϊκός λαός είναι από τους πρώτους που πίστεψαν στον Ιησού Χριστό, που υιοθέτησαν τις ιδέες του και που μετέφεραν το μήνυμά του σε όλο τον κόσμο. Μιλούν οι άνθρωποι αυτοί τη γλώσσα του Ιησού Χριστού. الاحتضار ونحتاج إلى معجزات لإنعاش هذا الشعب الأصيل في سوريا والتي أخذت اسمها منهم كسريان Nous sommes aujourd'hui un peuple qui vit à mort clinique. Είμαστε λαός που αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένα θαύμα για να ε, επανέλθει στη ζωή η Συρία, η χώρα που φέρει το όνομά μας.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 για να σας πούμε την ιστορία μας. Ωστόσο, ε, διωκόμαστε εδώ και χιλιάδες χρόνια, ε, ζούμε όμως ακόμη. Όπως είπε ο Χριστός ε, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, να προσέχετε τους όφης. وبالرغم من الدور الذي لعبه الكثير من الشخصيات السريانية في نهضة وتطور البلاد على كافة المستويات عانينا دائما من التهميش المقصود في الاعتراف بنا كشعب وهوية ولغة وذلك من كل الدساتير التي كتبت في فترات متلاحقة تمتد لعشرات من السنين وهذا Depuis la création de l'État syrien moderne, μετά τη δημιουργία του σύγχρονου κράτους της Συρίας, μετά την ανεξαρτησία, παρά το ρόλο που έπαιξαν οι άνθρωποι μας στην ανάπτυξη της χώρας, εμείς ε, οι χριστιανοί της ε, Συρίας ε, περιθωριοποιούμαστε, μας αρνούνται το εθνοτικό και γλωσσικό μας πλαίσιο. Εδώ και δεκαετίες συμβαίνει αυτό. وإنكار كل الهويات الأخرى ومنهم شعبنا السرياني واستعمال الترهيب والاعتقال لكل من ينشط نحو التكلم بهذه الخصوصيات ومحاولة إنعاشها. Tout cela s'est Tout cela a exprimé une même volonté des régimes successifs de supprimer les... Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν την βούληση των καθεστώτων να εξαφανίσουν τη μνήμη μας και να δημιουργήσουν μια ενιαία αραβική ιδέα για την περιοχή αυτή και να αρνηθούν την ύπαρξη κάθε άλλης εθνότητας με τρομοκρατία και με σύλληψη οποιοδήποτε ατόμου πρεσβεύει τις ιδέες αυτές. وأحيانا يطلق علينا أننا بقايا الصليبيين وفي أفضل الأحوال يطلق علينا الأقلية المسيحية Ce qui, ce qui a fait que la majorité des chrétiens de Syrie... Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι Σύριοι χριστιανοί ε, αρνούνται την ε, ταυτότητά τους ε, παρότι είμαστε οι αυτόχθονες ε, της Συρίας. Μας αποκαλούν ε, χριστιανούς Άραβες, ε, στην καλύτερη περίπτωση μας αποκαλούν χριστιανή, χριστιανική μειονότητα. Ναι. Le Parti de l'Union syriaque, dont je suis membre depuis sa création en 2005, το Ενωτικό Κόμμα της Συρίας από τη δημιουργία του το 2005 ε, συνενώνει τους ε, ανθρώπους του δικού μας λαού, του Αραμαϊκού, ε, και υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους. εάν οι άνθρωποι μας μπορούν ε, να απολάβουν των δικαιωμάτων τους, ε, θα μπορούν να συμμετέχουν και περισσότερο στις δημοκρατικές διαδικασίες. وغير ذلك هو النتيجة التي تحصل اليوم وهجرة أكثر من نصف مسيحي سوريا في ظل هذه أكثر من نصف مسيحي. Sinon, le seul résultat possible. Εάν όμως όχι, το μόνο πιθανό αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε και τώρα, ότι οι μισοί χριστιανοί έχουν φύγει από τη χώρα. Sachant que la migration chrétienne existait auparavant, mais elle se faisait en petit nombre. تم طرح مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية وكنا نحن من المؤسسين لها وذلك لأننا وجدناها ذات فكر يعترف بنا كشعب ودين ويحقق بين الجميع بمختلف القوميات والأديان. Έχουμε δει και στο παρελθόν ε, μετανάστευση των ε, χριστιανών. Η ιδέα είναι να έχουμε αυτόνομο δημοκρατικό κράτος. Euh, Θεωρήσαμε ότι κάτι τέτοιο θα μας επιτρέψει να ζούμε ως, δημοκρατική, ως θρησκευτική κοινότητα με ισότητα ανάμεσα σε όλες τις εθνοτικές ομάδες. Ce qui renforce la cohésion sociale, contrairement à ce qui était appliqué par les anciens régimes. Κάτι που θα οδηγήσει σε κοινωνική συνοχή σε αντίθεση με τα όσα ε, έχουν κάνει προηγούμενα καθεστώτα που προσπαθήσαν να διαιρέσουν ε, την ε, κοινωνία μας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 μπορούμε να ενώσουμε τις ε, δυνάμεις μας ε, και να αντισταθούμε σε ομάδες ε, όπως είναι το ΝΤΑΕΣ. Μας έχουν εξαφανίσει, μας έχουν εξορίσει από διάφορες περιφέρειες που έχουν καταλάβει. Επειδή είμαστε χριστιανοί, μπορεί να μας αποδυναμώσουν, δεν θα παραδοθούμε όμως, δεν θα εξαφανιστούμε ποτέ.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 κυβέρνησή μας ε, στην ε, αυτόνομη ε, διοίκησή μας. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχουμε διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις και έχουμε λάβει οικονομικά μέτρα για τους ανθρώπους μας. Την... Έχουμε κερδίσει την αυτονομία των ανθρώπων μας και έχουμε ενισχύσει το ρόλο των γυναικών. ونحاول أن نؤسس لسوريا جديدة تكون قائمة على إلغاء النظام المركزي الشوفيني وأعطاء دور للمناطق والأقاليم في إدارة شؤونها من خلال نظام لا مركزي ضمن وحدة سوريا Nous avons toujours essayé à travers notre projet d'être Πάντα προσπαθούσαμε να παρέχουμε λύσεις στη Συρία. Να δημιουργήσουμε μια νέα Συρία απειλαγμένη από τον κεντρικό σοβινισμό και όπου οι διάφορε ομάδε ε, να μπορούν να εφαρμόσουν τα δικά του συστήματα εντό μια ενωμένη Συρία. C'est vrai que nous avons eu des alliés dans notre guerre contre Daesh. Πράγματι, είχαμε συμμάχους ε, και είμαστε κατά του Daesh. Είχαμε συμμάχου σε την, το διεθνή συνασπισμό. Τώρα όμω βρισκόμαστε μόνοι, απομονωμένοι σε μια πολιτική σύγκρουση και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ πέρα σήμερα. وطموحات أغلب السوريين وخصوصا إننا نعاني وما, زل وما زلنا من الكثير من الأطراف السورية من التهميش لهويتنا وحقوقنا ونجد بأن أي دستور جديد في سوريا لا يتضمن فيه الاعتراف بنا كهوية شعب له حقوقه القومية والدينية والثقافية فهذا سيكون بمثابة الضربة القاضية لاستمرار وجودنا في بلدنا التاريخية سوريا Ce qui ne fait craindre qu'aucun changement véritable ne verra le jour dans... Δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κάποια πραγματική αλλαγή στη χώρα. Πολλές από τις πολλούς από τους διάφορους φορείς στη Συρία περιθωριοποιούν την ε, δική μας ταυτότητα. Δεν μας αναγνωρίζουν ε, ως ε, ξεχωριστό λαό με εθνοτικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά δικαιώματα. Αυτό όμως είναι μοιραίο χτύπημα στην ύπαρξή μας. التي تهدد وجودنا من قبل الكثير من القوى المحلية والإقليمية ونتعرض لحرب إبادة أمام أنظار جميع العالم لذلك نحن نطالب دائما بضرورة اهتمام العالم تجاه ما نتعرض له وكل ما نطلبه هو إيقاف كل الهجمات التي تحصل ضدنا كما نطالب بضرورة تطبيق الحظر الجوي لمناطق شمال وشرق سوريا Actuellement, dans le nord-est de la Syrie, nous nous retrouvons face à des menaces existentielles. Στα βορειοανατολικά της Συρίας αντιμετωπίζουμε υπαρξιακές απειλές ε, βρισκόμαστε σε πόλεμο με στόχο την εξαφάνισή μας και γι' αυτό θα σας παρακαλούσαμε να παρέμβετε εσείς για να σταματήσετε τις επιθέσεις εις βάρος των ανθρώπων μας. الضامن لمنع حصول إبادات جديدة على الشعب المسيحي وعموم المكونات الأخرى في المنطقة وسأذكر مثال واحد على ما أقول هو منطقة الخابور Cela va constituer une garantie pour qu'une nouvelle extermination αυτό θα αποτελέσει εγγύηση για να αποτραπεί η εξαφάνιση των χριστιανών της περιοχής. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, αυτό που συνέβη στο Χαμπούρ. هجوم عليها من قبل تنظيم داعش عام 2015 وحصل تهجير كامل لسكان هذه المنطقة كما أن داعش استطاع أن يخطف المئات منهم وأغلبهم من الأطفال والنساء وارتكبت جرائم بحق الكثيرين Dans la région de Khabour, euh, la région de Khabour pardon, était στο Χαπούρ. Ήταν ε, αποκλειστικά χριστιανικός ο πληθυσμός. Ε, το 2015 επιτέθηκε τον ΤΑΕΣ και ε, οι χριστιανοί αναγκάστηκαν να φύγουν. Έγιναν απαγωγές κυρίως γυναικών και παιδιών από την πλευρά του ΤΑΕΣ.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 στην ίδια περιοχή, αφού απελευθερώθηκε, επέστρεψαν κάποιοι από τους κατοίκους, ε, δέχτηκαν όμως εκ νέου απειλές από διάφορες ε, ακραίες μουσουλμανικές ομάδες, ε, που οδήγησε σε δεύτερη διαφυγή των ανθρώπων, χωρίς να λάβουν καμία βοήθεια από τον πολιτισμένο κόσμο. وكان Δυστυχώς ε, συνεχίζονται οι τραγωδίες αυτές. Ένας ιερέας και ο πατέρας του σκοτώθηκαν. Ε, είχαμε μία ε, έκρηξη κοντά στο Ραμίσλιο που ζω εγώ και ο γιο μου ήταν, ε, απήχε μόλι 100 μέτρα από το σημείο που έγινε η έκρηξη. Κλείνοντα ε, θα ήθελα... Θα θέλαμε να διατηρήσουμε την παρουσία των χριστιανών στην περιοχή αυτή και να ε, πετύχουμε σταθερότητα στην περιοχή.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 حيث من غير الممكن أن يتم استبعاد الإدارة الذاتية بكل مكوناتها من هذا الحدث المهم ولا بد أن ننقل ما قمنا به في مناطقنا على مستوى سوريا عامة وعبر دستورها الجديد Thank you. Il faut assurer une transi transition démocratique selon les décisions. Χρειάζεται να υπάρξει δημοκρατική μετάβαση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Θα πρέπει να έχουμε ένα δίκαιο και δημοκρατικό σύνταγμα που να διασφαλίζει τα δικαιώματα των χριστιανών ε, και να προστατεύει τον πολιτισμό και την γλώσσα μας. Θα πρέπει να είναι ένα σύνταγμα που να ε, μας καθιστά ίσους με όλους τους άλλους σύρους ε, για να υπάρξει ένα τέτοιο σύνταγμα θα πρέπει στην συνταγματική συνέλευση να υπάρξει ε, σωστή αντιπροσώπηση δεν ε, μπορούν να αποκλειστούν οι διάφορες περιφέρειες από μια τέτοια συνταγματική συνέλευση. Έχουμε δικαίωμα να ε, ε, εξηγήσουμε όλα όσα έχουμε κάνει στην περιοχή αυτή μέσω ενός νέου συντάγματος. Euh, λοιπόν, θα ακούσουμε κάποιους ομιλητές μετά από τα συγκλονιστικά πράγματα που πληροφορηθήκαμε. Ο λόγος στον Νατιό που είναι εισηγητής μας για θέματα Τουρκίας και από εκεί και πέρα θα δώσω το λόγο στον, στους, ε, ε στις πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα αυτό έχει συζητηθεί σε διάφορες επιτροπές, από τη σκοπιά που απασχολεί την κάθε επιτροπή βεβαίως Εμάς βεβαίως το θέμα μας απασχολεί κυρίως από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Τουρκία με την ε, εισβολή της επιδιώκει και μια δημογραφική αλλαγή. Δεν θέλει να επιστραφούν οι, ε, όλοι αυτοί που έχουν εκτοπιστεί στα μέρη τους, θέλουν να ανακατανεμηθούν μέσα στη Συριακή επικράτεια. Η Τουρκία λοιπόν θέλει ακόμη και να ιδρύσει νέες πόλεις και λέει ότι εγώ θα επιδιώξω αυτούς τους στόχους και αν δεν τα καταφέρω μπορεί να υπερβώ ακόμη και αυτούς τους ε, στόχους που είχα θέσει αρχικώς. Βεβαίως πρόκειται για μια κίνηση σε τεντωμένο σκηνή. Εμείς θα θέλαμε να βοηθήσουμε βεβαίως χωρίς ταυτόχρονα να ε, ενισχύσουμε την Τουρκία στα όσα παράνομα κάνει. Βλέπουμε την τελευταία περίοδο πραγματικά αποτρόπες πράξεις. Ε, σημαδεύονται σπίτια τη νύχτα. Πράγματα που έχουμε δει ε, και εδώ στην Ευρώπη, στην ιστορία της Ευρώπης. Πρόκειται για μια ευθεία απειλή κατά ανθρώπων και κάθε άνθρωπος έχει, έχει δικαίωμα να προστατεύεται από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους. Ε, όλοι οι άνθρωποι έχουν, ε, ε, καλύπτονται από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορεί κάποιες ομάδες να απειλούνται περισσότερο από άλλες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο βασικές μεταναστευτικές ροές. από την ε, βορειοανατολική ε, Συρία προς την Τουρκία και από τη δυτική Συρία προς την Τουρκία. Και ο Ερντογάν απαιτεί να λάβει χρήματα για την υποδοχή αυτών των ανθρώπων. Η διεθνής ε, αμνηστία ισχυρίζεται ότι πρόκειται για απάτη από πλευράς του Ερντογάν, διότι πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί που επιστρέφονται στη Συρία από την Τουρκία δεν γνωρίζουν πού θα, πού θα βρεθούν. Πολλές φορές συλλαμβάνονται ακόμη και στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και ε, ξαναβρίσκονται μέσα σε λίγες ώρες στη Συρία. Και η Τουρκία δεν κάνει τίποτα για να υποστηριχθούν και ε, οι άμαχοι θύματα των στρατιωτικών της επιχειρήσεων. θα έπρεπε κανονικά εγγύητη της διαδικασίας να είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Πρόσφατα, σε ακρόαση με την ΕΙΕΔ, ο κύριος Κουτέρες προσφέρθηκε ο ΙΕ να δράσει ως επόπτης της διαδικασίας. Εμείς ελπίσαμε ότι θα πρόκειται για μια συμβολή στην τελική συντριβή των ε, τζιχαντιστών. Αντιθέτως όμως, βλέπουμε η Τουρκία να συλλαμβάνει τζιχαντιστές, να τους βάζει σε αεροπλάνα και να τους στέλνει σε χώρες που δεν γνωρίζουν καν ε, ότι πρόκειται να υποδεχτούν ε, τέτοιους τζιχαντιστές. Ευχαριστώ πολύ. Ραφαέλ αν θέλεις διερμηνία προς τα γαλλικά μπορείς να βάλεις τα ακουστικά σου. Εγώ την ακούω. Ιζαμπέλ Βίσλα. Ευχαριστώ καταρχάς για όλες τις πληροφορίες που μας ε, παρήχατε. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα όσα ακούσαμε σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί είναι μια κατάσταση πραγματικά απεχθής από ανθρωπιστική σκοπιά. Και δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να είμαστε απλώς θεατές. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η Τουρκία είναι σε θέση να ελέγχει τους συμμάχους της και τα όσα εκείνοι κάνουν υπό την ηγεσία της Τουρκίας. Θα ήθελα να μα πείτε περισσότερα στοιχεία σε σχέση με αυτό. Επιπλέον, στην αρχή της τοποθέτησή σα, των παρουσιάσεων σα, ακούσαμε διάφορα στοιχεία αριθμητικά όσον αφορά τους Κούρδους, τους κουρδικούς πληθυσμού που εγκαταλείπουν τις ε, ε, εστίες τους. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία συνεχίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε και αν ναι, προς τα πού πηγαίνουν κατευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι η διάκριση που περιγράψατε, οι διακρίση που διαγράψατε μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι αυτή η σύγκρουση ε, στην οποία συμμετέχουν η Τουρκία, ο Ασάντ, η Ρωσία ε, φαίνεται ότι είναι κάτι που δεν θα ε, λάβει τέλος σύντομα. Αναφερθήκατε και στους τζιχαντιστές και αναρωτιέμαι μήπως όλοι οι τζιχαντιστές βρίσκονταν εντός αυτής της επικράτειας που ε, ελέγχει η Τουρκία. Και αν ναι, πόσοι είναι. Και επίσης, έχετε διερευνήσει άλλες ε, λύσεις που θα μπορούσαν να δοθούν. Έχει ακουστεί η ιδέα της ε, δημιουργίας ε, ενός διεθνούς δικαστηρίου. Οργανώνεται κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Και Βεβαίω είμαι πάντοτε ιδιαίτερα περιχαρής όταν βλέπω γυναίκες να αναλαμβάνουν ηγετικέ ε, πολιτικές θέσεις και να μεταφέρουν τα μηνύματά τους. Πρέπει να πω ότι δεν έχω χάσει ακόμη την ελπίδα ότι είναι ε, εφικτή η συμβίωση όλων αυτών των πληθυσμών. Σοσιαλιστές η κυρία Ίντς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές ε, για τη σημαντική δουλειά που κάνουν και που ανταλλάσσουν μαζί μας ε, τις απόψεις τους ε, και τις εμπειρίες τους. Κλιμακώνεται η κατάσταση κάθε μέρα, όλο και περισσότερο. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, τρομοκρατούνται άνθρωποι από διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως εξηγήσατε. Και δυστυχώς ακόμη και από ε, τρομοκρατικές ε, οργανώσεις υπό την προστασία της Τουρκίας ή που έχουν την ευλογία της Τουρκίας. Για να έχουμε λοιπόν, ε, θέλουμε μία μακροπρόθεσμη πολιτική λύση και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανη για ε, το ψήφισμα που υιοθέτησε πριν δύο εβδομάδες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει με βάση αυτό το ψήφισμα και επίσης το Συμβούλιο να ε, πάρει σύντομα θέση ακολουθώντας τη θέση του Κοινοβουλίου, διότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για να μην χάσουν άλλοι άνθρωποι τη ζωή τους. Δεν επιτρέπεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Από τη μία λοιπόν θέλουμε πολιτική λύση, μία άμεση ε, πολιτική λύση και μία μακροπρόθεσμη πολιτική λύση. Το άλλο θέμα όμως είναι και η επίγουσα ανάγκη για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Γι' αυτό έχω δύο ερωτήσεις προς και τους τρεις ομιλητές. Πρώτον, ποιες οργανώσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή Ροζάβα. Δεύτερον, ποιες είναι οι πιο επίγουσες ανάγκες και ποιοι είναι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι να παράσχουμε ανθρωπιστική βοήθεια για να φτάσει στους ανθρώπους. Διότι γνωρίζω κάποιες χώρες που έχουν λάβει απόφαση αύξησης της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την περιοχή δεν έχουν βρει ακόμη όμως αποτελεσματικούς τρόπους να είναι αποτελεσματική αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας παρακαλούσα να συντομεύετε τις παρεμβάσεις σας για να προλάβουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις των ομιλητών μας. Ε, Ερωτήσεις έχω. Καταρχάς προς την κυρία Κορία. Γνωρίζετε εάν οι Τούρκοι θέλουν να αποχωρήσουν οι χριστιανοί από την περιοχή αυτή που καταλαμβάνουν αυτή τη στιγμή. όπως επιθυμούν για τους Κούρδους. Δεύτερον, εάν πράγματι ισχύει αυτό, πράγμα που από ό,τι φαίνεται ισχύει, Έχετε κάποια άλλη λύση να προτείνετε ε, πέρα από αυτό που έκαναν οι Κούρδοι, να ζητήσετε δηλαδή από το καθεστώς Ασάντ να σας υπερασπιστεί. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πιερίνη Πολύ χαίρομαι που σας ε, βλέπω εδώ. Πολύ καιρό είχα να σας δω. Πιστεύετε ότι οι Σύριοι πρόσφυγες πράγματι θέλουν να εγκαταλείψουν ήδη αύριο την ε, Τουρκία. ότι θα φεύγανε αύριο από την Τουρκία αν μπορούσαν, ε, διότι θα επιστρέψουν σε πολύ δύσκολες ε, συνθήκες, επικίνδυνες συνθήκες. Η ζωή στην Τουρκία μπορεί να μην είναι ρότινη, αλλά δεν βρίσκονται υπό απειλή 24 ώρες το 24 ώρες τα μέρες την εβδομάδα. Η κυρία Λάνια Ζήπεν, παρακαλώ. Θα μιλήσω γερμανικά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ε, τη συζήγηση σας. Ε, απελπισία με πιάνει με αυτά που ακούω. Από το ξέσπασμα του πολέμου το νιώθω αυτό. Η Τουρκία ε, και άλλοι βλέπουμε τον Τάις να γίνεται όλο και πιο ισχυρό στην περιοχή. Ο Ερτογάν γιατί το θέλει αυτό, διότι έχει έτσι μια ανταγωνιστική δύναμη την οποία δεν μπορεί να ε, ε, ελέγξει. Μπορεί όλο αυτό να φαίνεται πολύ πρακτικό και το λέω αυτό έτσι με, το λέω χοντρά, αλλά θα έχουμε έτσι έναν, θα έχει ο Ερντογάν έναν ανταγωνιστή τον οποίο δεν μπορεί να ελέγξει. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση και ακούσαμε ότι ο Ερντογάν και ο Πούτιν και ο Ασάντ Ε, θέλουν να μοιράσουν τη χώρα όπως τους βολεύει. Ε, το Ντάις έχει να παίξει και εδώ ρόλο. Και ποια είναι η αντίδραση μέχρι τώρα από τον Ασάντ. Θα μπορούσε να πει κανείς ηρωνικά ότι ο Ασάντ δεν έχει πολλά να πει ακόμη. Ο Πούτιν αποφασίζει, αλλά πώς έχει η κατάσταση εντός της ε, κυβέρνησης της Συρίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές μας για την παρουσία τους εδώ, ιδίως, της κυρίας, ιδίως την κυρία Κορέα. Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επίθεση ε, ήταν πραγματικά ντροπιαστική. καθώς ανεστάλησαν οι προμήθειες οπλικών συστημάτων προς την Τουρκία και λοιπά. Αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει είναι να ανασταλούν οι χρηματοδοτήσεις προς την Τουρκία ε, της, και στο πλαίσιο των, ε, της ε, προενταξιακής της πορείας. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει. Ξέρουμε τι θέλει να κάνει ο ε, Ερντογάν. Θέλει να εξαφανίσει τους χριστιανούς από τη Μέση Ανατολή. Πριν από 10 χρόνια ζούσαν 3 εκατομμύρια χριστιανοί ε, στην ε, Μέση Ανατολή. Το Σάββατο ε, ήμουν σε μια εκδήλωση μιας μη κυβερνητική οργάνωση στην Ουτρέχτη και εκεί ανακοινώθηκε ότι πλέον οι χριστιανοί που ζουν στη Μέση Ανατολή ανέρχονται σε 250.000. Γιατί, γιατί τους συνέτριψε ο Ερντογάν και ο πόλεμος. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι ή πλέον είναι πολύ αργά. Και ε, σπαταλήσαμε όλο μας το χρόνο μιλώντας εδώ σε διάφορα φόρουμ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Σάντος, θα ήθελα να απευθύνω ένα ερώτημα στον δημοσιογράφο που βρίσκεται στη Συρία. Μιλήσατε για τη χρήση οπλικών συστημάτων που έχουν την ε, προέλευσή τους από την Ευρώπη. Που ευρωπαϊκές χώρες δηλαδή έχουν προμηθεύσει την Τουρκία με αυτά τα οπλικά συστήματα. Έχετε συγκεκριμένες πληροφορίες για το ποιε ε, χώρες είναι αυτές που έχουν προμηθεύσει τον τουρκικό στρατό με οπλικά συστήματα. Όταν, όταν λέω ε, πληροφορίες δεν αναφέρομαι σε, φήμες. Αναφέρομαι σε συγκεκριμένες αξιόπιστες πληροφορίες για το από πού προέρχονται ε, αυτά τα οπλικά συστήματα, από ποιες ευρωπαϊκές χώρες. Ο κύριος... Ο κύριος Μπένιον, ναι, ευχαριστώ. Πριν τη συζήτηση που είχαμε στο Στρασβούργο πάνω στο θέμα αυτό, είχα μια συνάντηση με τον Τούρκο πρέσβη, που με ενημέρωσε ότι αυτή η περιοχή στα βόρειο-ανατολικά της ε, Συρίας ε, δεν είναι περιοχή Κούρδων ή ε, χριστιανών ε, είναι κατά 80% Αραβικοί. Αυτό ε, εμένα μου έκανε το συναγερμό να χτυπάει, διότι τι γίνεται εδώ. Υπάρχει συνωμοσία για να μεταφέρουμε τους Άραβες πρόσφυγες στην Τουρκία να πάνε στην περιοχή αυτή, ακόμα και αν δεν προέρχονται από αυτήν. Και ε, έθεσα αυτά τα ερωτήματα στην ΑΦΕΤ την προηγούμενη ε, εβδομάδα χωρίς να λάβω καμία απάντηση. Νομίζω ότι ήδη έχουμε την ε, απάντηση. Πρόκειται πράγματι για συνωμοσία ώστε να υπάρξει ανταλλαγή πληθυσμού και να πάνε εκεί άνθρωποι από άλλα μέρη της Συρίας που αυτή τη στιγμή είναι πρόσφυγες στην Τουρκία. Και αυτό είναι κοινικός οπορτουνισμός την Παρασκευή θα συναντηθώ με ανθρώπους, ε, ε, ε, με Κούρδους και θα ήταν χρήσιμο να μου πείτε Ε, μάλλον με το κόμμα του Ερντογάν έχω συνάντηση. Ε, θα ήθελα πολύ να μου πείτε πόσο να του πιέσω. Πάντα νομίζω ότι είναι χρήσιμο να έχουμε συναντήσει με τους ανθρώπους αυτούς. Ε, Πάντω φαίνεται να είναι σωστέ οι αρχικέ μου υποψίες. Πείτε μου σας παρακαλώ τι να πω στο κόμμα αυτό την Παρασκευή όταν συναντηθώ μαζί του. Η Julie Ward. Σας ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι που έχασα την εισήγησή σας, ε, αλλά βρίσκομαι εδώ διότι είχα σε επαφές με ανθρώπους ε, στην ε, Ροζάβα. Υγήθηκα μιας αποστολή γυναικών εκεί πέρσι και πραγματικά με ταράζει πολύ το να βλέπω τον χάρτη διότι πήγα σε πολλά τέτοια μέρη και γνωρίζω ότι άνθρωποι που συνάντησα μπορεί να έχουν ήδη τραυματιστεί ή σκοτωθεί. Ενώ ήμουν ικανοποιημένη με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν νομίζω ότι ε, τονίσαμε αρκετά την δημοκρατική επανάσταση στη Ροζάβα και τον τρόπο που ενδυνάμωσε τις γυναίκες να ανοικοδομήσουν την κοινωνία, όχι πρακτικά, ε, λίθο προς λίθο, αλλά να δημιουργήσουν νέα οικονομικά ε, πρότυπα. Είδαμε το χωριό γυναικών που επισκέφτηκα, να, όπου υπάρχει ένα πρότυπο δημοκρατίας που ε, σέβεται την ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Δεν ήταν ε, δυνατόν να το συμπεριλάβουμε αυτό στο ψήφισμα. Ξέρω ότι η Πατρίσια Τόγια έκανε εξαιρετική δουλειά, άκουσε τις πληροφορίες που ε, είχα λάβει απευθεία από Διεθνή Οργανισμό Γυναικών. Ε, ήμουν απλά διεύλο, αλλά δυστυχώς αυτό δεν πέρασε από την Ολομέλεια. Νομίζω ότι Έχουμε σημαντικό πρόβλημα όταν δεν αναγνωρίζουν οι άνθρωποι αυτά που έχουν γίνει επί τόπου τα τελευταία χρόνια. Και το λέω διότι τα είδα εγώ αυτά με τα ίδια μου τα μάτια. Πολλοί άνθρωποι μιλούν για τα πράγματα αυτά εδώ. Δεν, δεν τα είδαν όμως με τα ίδια του τα μάτια. Εγώ θα ήθελα να είμαστε πολύ πιο ε, τολμηροί, θαραλέοι και πολύ πιο ειλικρινεί όσον αφορά την αξιολόγησή μα των όσων συνέβησαν εκεί τα τελευταία χρόνια. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Η κυρία Νόημαν. Ένα ερώτημα κυρίω για τον κύριο Περίνη. Όταν εξετάζουμε την κατάσταση των ε, Κούρδων προσφύγων που είναι εγκλωβισμένοι, εγώ βρέθηκα στην περιοχή ε, πριν από μια εβδομάδα και οι Ιρακινοί ε, εμποδίζουν τους Κούρδους να εισέλθουν στο ε, έδαφος της χώρας για να μην υπάρξει δημογραφική αλλίωση. Από την άλλη πλευρά, από ανθρωπιστική σκοπιά, είναι η μόνη λύση που μπορεί να δοθεί για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω εσείς ποια, είναι, ποια πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είναι η λύση. Για τη συνταγματική συνέλευση. Ξέρω ότι οι ΙΠΑ πίεσαν να συμμετάσχουν οι ε, αντιπολιτευόμενες δυνάμεις. Οι Κούρδοι δεν συμμετέχουν. Δεν ξέρω ποια είναι ε, η αίσθησή σας σε σχέση με αυτό. Και θέλω συγκεκριμένα να μου πείτε στις διαπραγματεύσεις αυτές αν παίζουν κάποιο ρόλο τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως η ε, κατάργηση της ασυλίας. Επίσης, η Σύνοδος ε, Υπουργών Εξωτερικών επέβαλε σήμερα κυρώσει στην Τουρκία για την εξόρυξη πετρελαίου στη Μεσόγειο, αλλά δεν κατάφερε να επιβάλλει αντίστοιχε κυρώσει για την κατάσταση και τα όσα έχει διαπράξει η Τουρκία στη Συρία. Η κυρία Στρίκ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους ε, ομιλητέ μα για την εξαιρετική παρουσίαση της κατάσταση στην Βορειοανατολική Συρία. Για την κατάσταση των Κούρδων και των ε, χριστιανικών ε, πληθυσμών στη Συρία, τα πράγματα ήταν σαφή, περιγράφηκαν με κάθε σαφήνεια βεβαίως και ε, είναι πολύ ανησυχητικά τα πράγματα. Θα ήθελα να μου πείτε και οι δύο τι πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κάνει αυτή τη στιγμή τι χρειάζεστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μπορέσετε να προστατεύσετε τα δικαιώματά σας, διότι είναι σαφές ότι βρίσκονται ε, ε υποκαθεστώς επίθεσης. Ε, και ε, είναι σαφές ότι για το ψήφισμα και το εμπάργκο πώληση ε, οπλικών συστημάτων δεν έχουν αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε για την προστασία των χριστιανικών και κουρδικών πληθυσμών στο πλαίσιο αυτή τη ειρηνευτική διαδικασία. Για τον κύριο Περίνη, θα ήθελα να τονίσω κι εγώ ότι ο ρόλο Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν περιορισμένο και πλέον φαίνεται να περιορίζεται ακόμα περισσότερο λόγω της κατάστασης έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, κάτι που μας οδηγεί στο να αναρωτηθούμε στο τι τελικά μπορούμε πια να κάνουμε. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να αποκαταστήσουμε κάποιες γέφυρες με τους Ρώσους προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα των πληθυσμών εκεί προστατεύονται επαρκώς. Όσον αφορά τις επιστροφές και τις πιθανές επιστροφές προσφύγων, εγώ συμφωνώ. Αυτό θα ήταν παραβίαση της ε, ε σύμβασης για τα δικαιώματα των ε, προσφύγων, αν γίνουν τέτοιες επιστροφές αυτή τη στιγμή ε, και πώς, ποιος θα παρακολουθούσε κιόλας μια τέτοια διαδικασία. Κατά τη γνώμη σας, αν γίνει μια τέτοια επιστροφή μαζική, Ποιο θα πρέπει να, είναι, να δρά ω εποπτική αρχή και τι θα έπρεπε και θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για τι μειοψηφίε και ορθώ γιατί είναι στόχοι. Και είπαμε για του Κούρδου από πλευρά των ε, Τούρκων αλλά γενικά θίγονται και οι Χριστιανοί. Τι γίνεται με τους ε, Σύρους πέραν χριστιανών και πέραν ε, Κούρδων μήπως θα πρέπει και εκεί να δούμε τι γίνεται, τι γίνεται με τους πολίτες, με τους ε, άμαχους Σύρους. Αυτοί είναι τα μεγάλα θύματα αυτού του πολέμου ευθύ εξ αρχή. Ίσως ο Ραφαήλ μπορεί να μας τα πει αυτά. Ο Μάρκ γιατί θα πρέπει να φύγει. Εσείς και μετά ο Ραφαήλ και μετά εσείς κυρία θα κλείσετε. Όσον αφορά ε, αυτές τις απελάσεις τζιχαντιστών είναι προφανές ότι όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα χάος. Ο, ο πρώτος σήμερα το πρωί ένας Αμερικανός ε, διώχτηκε και έχετε και στο ίντερνετ τι φωτογραφίες του και βρέθηκε σε αυτή τη ζώνη προστασία μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία, αυτό είναι μόνο του εκεί στο δρόμο. Δεν ξέρω αν έχει τι βαλίτσε του, οι, οι Έλληνες αρνούνται να τον υποδεχτούν, οι Τούρκοι αρνούνται να τον πάρουν πίσω. Έτσι είναι η κατάσταση και φυσικά τα πράγματα θα έχουν και άλλε εξελίξει. Είπαμε, αυτό είναι το σχήμα. Ε, ακριβώ όπω έγινε και μεταξύ Γαλλία και Τουρκία. Πάρα πολύ δυσάρεστα όλα αυτά. Ε, όλα αυτά είναι λάθο, όλα αυτά είναι φάουλ. Ει βάρο των χρόνων όπου είχαν ηθαγένεια αυτή. οι τζιγαντιστέ όσον αφορά την επιστροφή από την Τουρκία προ τη Συρία. Ε, σήμερα τα πράγματα είναι στο χειρότερο δυνατό σενάριο ε, σας είπα όλα τα προβλήματα και εσείς μας αναφέρατε και το, το, μόνο σχήμα το διαχειρίσιμο είναι ε, να πάνε τα πράγματα στο βήμα του ΟΗΕ, να βρεθεί εκεί πολιτική λύση για τη Συρία και υπό την πίεση της Ένωσης η Ρωσία να βοηθήσει να λειτουργήσει ο μηχανισμός και να γίνει τέτοιου είδους διευθέτηση και έτσι να μπορέσουμε να καθιερώσουμε κάποιο σχήμα για τους Κούρδους της Συρίας. Όπως είπαμε από το 12 δεν μπορούν να έχουν κάνει ταυτότητα να και εάν κλείσει συμφωνία μπορεί να πάρει ένα-δύο χρόνια ή παραπάνω και έτσι, αν έχουμε και αυτή τη δύναμη για να εγγυηθεί την τήρηση αυτών των συμφωνιών, τότε ίσως να έχουμε μια επιστροφή ε, μέχρι τότε. Αυτά δεν ξέρω αν μπορούμε να πείσουμε τους Σύρους. Ε, καλά, όχι τα, τα παιδιά που δεν καταλαβαίνουν, αλλά τους Σύρους της Κωνσταντινούπολης ή της Άγκυρας ή των Αδάνων να επιστρέψουν στη χώρα τους ε, αλλά όχι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Ξέρουν, ξέρουν τι γίνεται καθεστώς Σάσαντ και δεν θέλουν να γυρίσουν. Πολλοί από αυτούς έχουν ενταχθεί στην ε, ε, τουρκική οικονομία, σε τουρκικές εταιρείε, με τη βοήθεια της και αλλιώς της Ένωσης, οπότε δεν είναι σίγουρο κάνω ότι οι εργοδότες θέλουν να τους αφήσουν να φύγουν. Οπότε η κατάσταση αυτή είναι πολύ άνηση Έχουμε διάφορες εκθέσεις όπως ε, το International Crisis που περιγράφει πώς είναι η κατάσταση ιδίως στον Νοτιοανατολική Τουρκία σε σχέση με τον τουρκικό πληθυσμό γιατί εκεί έχουμε μεγάλη πυκνότητα πληθυσμό, ε, σε σχέση με τους πρόσφυγες αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα για αυτά τα 3,6 ε, ε, εκατομμύρια που λένε Τώρα, δύο λόγια ακόμα για το τι πρέπει να κάνει η Ένωση. Εάν υπάρξει κυβέρνηση, θα πρέπει το Συμβούλιο να αποφασίσει να μπει σε κίνηση η Ευρωπαϊκή Δημοπλατεία. Είχαμε τρεις διασκέψεις πέρσι για την ε, Συρία που έκανε η κυρία Μογκερίνη. Αγνοήθηκαν όλα αυτά από τα κράτη-μέλη που προτιμούν τις συναντήσεις κορυφής με Πούτιν και Ερντογάν. Γαλλία και Γερμανία. Οπότε η συνθήκη της Λισαβόνας λέει κάποια πράγματα που τα οποία δεν τηρήθηκαν. Λέει ότι θα πρέπει όλοι να ε, δρούμε μαζί. Ξέρετε γιατί δεν τηρήθηκαν αυτά. Αλλά Εάν δεν κινηθεί ε, όλη μαζί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα κάνουμε τίποτα. Ραφαήλ, έχει τρία λεπτά, μάλιστα. προσπαθώ να σα τα πω γρήγορα. Όσον αφορά τώρα τι ομάδε που ελέγχει η Τουρκία, η άλλη μια φορά ανέλαβε ευθύνη για την ε, δολοφονία των ε, αμάχων η Τουρκία. Δεν έχει πρόβλημα και την ε, ηγέτησα των Κούρδων επίσης. Ε, βεβαίως και δρούν με χαοτικό τρόπο αυτές οι ομάδες, κάνουν ό,τι θέλουν, πάνε όπου θέλουν και δεν υπάρχει καμία κύρωση για όσα κάνουν. Ξέρει πάρα πολύ καλά η Τουρκία ότι αυτά την ωφελούν, τα ελέγχει. Τώρα όσον αφορά τις ε, τη μετακίνηση του πληθυσμού. Έχουμε 30.000 κόσμο που έχει φύγει μετά την επίθεση στη Ράκα και στο Ιράκ. Τώρα εδώ έχουμε τρει ΜΚΟ που εργάζουν, την Βασόρ, ε, τον, κόκκινο, τον Ερυθρό Σταυρό, ένα, ε, ένα γερμανικό επίσης και η Βασόρ είναι ε, ο Ερυθρό Σταυρός των Κούρδων και νομίζω ότι αυτοί ε, συνεργάζονται με την Ευασόρ για να βοηθήσουν. Τώρα, όσον αφορά τον ε, Άσαντ, θέλει να επιστρέψει τα πράγματα όπως ήταν πριν τον πόλεμο. Αυτή είναι η θέση του, η πάγια. Ε, και βέβαια δεν κρύβει το ότι ο στόχος του είναι η υποταγή της περιοχής όσο μπορεί. Τώρα όσον αφορά τα όπλα αυτά, ε, ε, έχουμε φωτογραφίες, έχουμε βίντεο για τα Leopard, σας το επιβεβαιώνω και αν θέλετε να σας πω και άλλα στοιχεία να σας τα στείλω. Όποτε θέλετε μπορεί να έρθετε σε επαφή μαζί μου και έτσι θα έχετε αποδείξεις για τα ε, Leopard αλλά και για άλλα θέματα που τυχόν σας ενδιαφέρουν. Επίσης όσον αφορά τους υπόλοιπους ε, μη Κούρδους, μη χριστιανούς. Είναι φυσικά κατά και οι Άραβες, κατά της επίθεσης της τουρκικής. Παντού, στη Ράκα, σε όλη τη Βόρεια Συρία έχω μιλήσει με Άραβες. Οι περισσότεροι λένε όχι, μόνο οι τζιχαντιστές, μόνο οι Νταές είναι υπέρ. Και αυτοί βγαίνουν στον τύπο και λένε ναι, ναι, ναι, περιμένουμε. Περιμένουμε την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Αυτοί το λένε. Ε, αυτό είναι, είναι τόσο, τόσο ηρωνικό, τόσο αστείο. Ε, οι Άραβες είναι κατά. Ε, έχουν χτυπηθεί, έχουν πάθει από το Ισλαμικό κράτος και από τους Τούρκους. Και στη Ράκα, ακριβώς. Αυτά πρεσβεύουν. Άρα είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε γι' αυτό. Οπότε, εν κατακλείδη, Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος. Υπάρχουν ε, συμφωνίες ελεύθερης, ε, ε, ελευθέρων ανταλλαγών μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης. Ας τις εκμεταλλευτούμε. Δεν είναι να, καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα. Άλλωστε είναι και όλες οι εξαγωγές οι Τουρκίες προς την Ευρώπη. Κάντε κάτι, μπλοκάρετε εδώ για να κάτσει να προβληματιστεί ο Ερντογάν. να σταματήσουν οι πτήσεις των Τούρκων και μου είπε ο Κούρδο ε, Υπουργό, το πρόβλημα είναι οι αεροπορικέ επιθέσει. Εάν δεν μπορούσαν οι Τούρκοι να επιχειρήσουν με τα αεροπλάνα, τότε δεν θα μπορούσαν να προωθηθούν τα τουρκικά στατεύματα και οι ομάδες που βοηθούν τους Τούρκους. Οπότε, θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, να ζοριστεί οικονομικά η Τουρκία, να σταματήσουν όλα αυτά. Αυτή είναι όλη την επίθεση που άλλωστε κοστίζει τόσο πολύ. Πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν μπορούν, δεν μπορούν να μείνουν πολύ καιρό χωρί να ξοδέψουν ένα σωρό λεφτά. Επομένω, ε, θα πρέπει κάπω να κάνουμε για να, το, να του αδειάσει το πορτοφόλι. Ραφαήλ, σε ευχαριστούμε, λέει πρόεδρο. Στο μέλλον θα είμαστε σε επαφή. Και την τελευταία κυρία Ναζίρα.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 των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο Ερντογάν είπε ότι δεν έχει ε, σκοπό να αλλάξει κάτι όσον αφορά τις χριστιανικές κοινότητες στη Συρία. Αν κοιτάξτε το χάρτη όμως θα διαπιστώσετε ότι η περιοχή που θέλουν να καλύψουν είναι αυτή ακριβώς όπου βρίσκονται τα χωριά των χριστιανών. Ιδιαίτερα το Ντάλτμερ και το Χαμπούρ έχουν ε, δεχτεί επιθέσεις. Πρόκειται για χριστιανικές περιοχές. وسهل نينوي بوضع كانوا وضعوا حرف النون على منازل المسيحيين لأخذها للجهاديين واليوم نفس الأسلوب برأس العين وبهذه المناطق يتم أحد وضع علامات على منازل المسيحية لأخذها للجهادين الموجودين هنا. Donc les groupes radicaux euh, qui sont présents maintenant dans le nord de la Syrie utilisent les mêmes méthodes que, le, que Daesh. Οι ε, ριζοσπαστικέ ομάδε στην Συρία χρησιμοποιούν τι ίδιε μεθόδου με τον Daesh και το ISIS. Σημαδεύουν τα σπίτια των χριστιανών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 فنحن معرضين جميعا هذه المكونات بهذه المناطق لاستهداف التركي ومن ممارسات القوات أو, أو الجروبات المسلحه المتطرفه التي تدخل هذه المناطق Donc la violence que, que, que la violence qu'il s'exerce maintenant dans le nord de la Syrie est aveugle. Il fait... Η βία στα βόρεια της Συρίας είναι τυφλή, δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε χριστιανούς Άραβες ή Κούρδους. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν δίπλα-δίπλα. Δεν γίνονται λοιπόν διακρίσεις, όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουν ε, τους βομβαρδισμούς. Οι βομβαρδισμοί γίνονται τυφλά. هدف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 Έτσι, αναγκάζονται οι άνθρωποι μας να εγκαταλείψουν ε, τις εκτάσεις αυτές. Ε, είναι σαφής ο στόχος του Ερτογάν η δημογραφική, η δημογραφική αλλαγή. Και μάλιστα στο σύνολο της ε, μεσογειακής περιοχής μέχρι τη Μοσούλη θέλουν να ξαναελέγξουν τις πρώην Οθωμανικές περιοχές. اليوم وكنا نحن وافقنا على دخول قوات النظام لحماية الحدود لأن هذه من واجبه. Donc, euh, concernant la deuxième question. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, και εμείς αναρωτιόμαστε, είναι σε θέση το καθεστώς να μας προστατεύσει? Υπάρχει τώρα η Ρωσοτουρκική συμφωνία και έτσι υπάρχει υποχρέωση προστασία μα, αλλά αυτό ζητάμε εδώ και πολύ καιρό. Euh, Αναζητούμε απεγνωσμένα πολιτική λύση. Το καθεστώς όμως δεν θα μας επιτρέψει να απολαύουμε των δικαιωμάτων μας. Δεν θέλει να αναγνωρίσει τα δικαιώματά μας και δεν θέλει να επιστρέψουμε στο στάτους quo που επικρατούσε πριν. Εμείς αυτό θέλουμε απλά. ولكن نحن لن نقبل بهذا الشيء فنحن نسعى لحل سياسي ديمقراطي لنثبت حقوق كل المكونات كرد عرب سوريان الجميع يكون حقوقهم موجودة بدستور ديمقراطي يضمن حقوق الكل Donc il veut revenir à 2011 Θέλουν λοιπόν να επανέλθουν στο 2011 να ελέγχουν το σύνολο της έκτασης ε, της ε, Συρίας. Εμείς όμως δεν θα το δεχτούμε αυτό. Θέλουμε μια πολιτική, δημοκρατική λύση που να επιτρέπει σε όλους ε, να ασκούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα. Σε Σύριους, Χριστιανούς, Άραβες... Je sais que pas Γνωρίζω ότι δεν είχα πολύ χρόνο να σας τα εξηγήσω όλα αυτά. Έχουμε όμως μια παροιμία. L'eau Όποιος έχει τα χέρια του στο νερό δεν καταλαβαίνει τη θέση αυτού που έχει τα χέρια του στη φωτιά. لحل سياسي ودفع أن يكون إيقاف هذا الهجوم ويكون وجود عقوبات على أردوغان وعلى حكومة تركيا. Donc, euh, le temps passe et c'est nous qui perdons notre... Ο χρόνος περνά. Χάνουμε τους ανθρώπους μας, ε, βρίσκονται στην εξορία, χάνουμε την ιστορία μας, χάνουμε τα εδάφη μας και γι' αυτό θέλουμε επιγόντως μια πολιτική λύση. Θα θέλαμε να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία. يوميا تفجيرات بأحيائنا وبين بيوتنا وأيضا قتل الكهنة المسيحيين وقتل كل المكونات الموجودة فيجب أن يقف عن هذه الممارسات Il faut surtout arrêter ces tentatives de, de, de réanimer Daesh, de le ramener à la vie. Χρειαζόμαστε Χρειάζεται να σταματήσουμε τις προσπάθειες ε, να ε, αναβιώσει το ISIS. Πρέπει να σταματήσουν οι επιθέσεις του ISIS, διότι δολοφονούν τους, πολιτικές, τους πολιτικούς μας ηγέτες. Θέλουμε να σταματήσουν όλα αυτά. J'ai difficile à euh, Δυσκολεύομαι να εκφράσω. Νιώθω μεγάλη συγκίνηση, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε τους ε, λαούς ε, της ε, Συρίας να μείνουν εκεί. Η Συρία δεν πρέπει να χάσει αυτό το σημαντικό στοιχείο των αυτοχθόνων της περιοχής. Σούρια. لأن يجب أن تكون مرخصة أو تدخل عن طريق دمشق الحكومة السورية وهناك صعوبة إلى مناطقنا euh, Όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις ΜΚΟ να δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. Πριν ε, καταφτάσουν πρέπει να ζητήσουν έγκριση από το καθεστώς το καθεστώ δεν δίνει τέτοιες εξουσιοδοτήσει. Euh. Πρέπει να βρούμε τρόπο να αποσταλεί ανθρωπιστική βοήθεια κατευθείαν στα νοτιοανατολικά τη Συρίας σε συνεργασία με ΜΚΟ που ήδη βρίσκονται εκεί. Ιδιαίτερα ε, η κουρδική ερυθρά Έλληνο θα πρέπει να καταφτάσει στην περιοχή. Σας ευχαριστώ. Euh, Για πάρα πολύ λίγη ώρα, μια που έχουμε καθίσει τους πολύ να πάρει το λόγο εταιρεία Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την έναρξη της ε, σύγκρουσης στη Συρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει διαρκώς ε, την ανησυχία της για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη χρήση βίας, όπως είναι οι εξοδικαστικές ε, δολοφονίες πολιτών, τα βασανιστήρια, η χρήση χημικών όπλων και η καταστροφή των συριακών υποδομών. Με αυτόν τον τρόπο εκφράσαμε τις απόψεις μας ε, σε όλα τα διεθνή φόρα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Συνεχίζουμε να καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να συμβάλλουν στην προστασία των αμάχων και των εργαζομένων των ε, ανθρωπιστικών οργανώσεων. Πρόσφατα, ε, μετά την μονομερή τουρκική εισβολή στην ε, βορειοανατολική ε, Συρία. Καταγράφηκαν πολλές παραβιάσεις ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολλές εκ των οποίων διεπράχθησαν από Σύριους οι οποίοι είναι σύμμαχοι των τουρκικών στρατευμάτων. Κάποιες από αυτές τις αδικοπραξίες, όπως είναι οι δολοφονίες αμάχων, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ακόμη και εγκλήματα πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδικάσει επανειλημμένω τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην ε, βορειοανατολική Συρία. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στην ε, θέση ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη και λογοδοσία. Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε την ανεξάρτητη, υποστηρίξαμε μάλλον την ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα COI το 2011. Επίσης έχουμε ε, ε, τονίσει επαλληλειμμένως ότι τα μέλη αυτή τη Επιτροπής θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στη Συρία. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να χρηματοδοτεί όλους τους ε, μηχανισμούς λογοδοσίας, όπως είναι το Διεθνές Γραφείο Αγνοουμένων τον ε, Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και την ε, Επιτροπή Λογοδοσίας που ε, διερευνά τις υποθέσεις που σχετίζονται με όλες τις πλευρές της σύγκρουσης. Αυτά είναι τα ζητήματα που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσά που ανέρχονται σε 16,6 εκατομμύρια ευρώ. Σε σχέση με τις μελλοντικέ επιστροφές, Αυτέ θα πρέπει να γίνουν με βάση τα διεθνή κριτήρια που έχει καθορίσει η αρμοστία για του πρόσφυγες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ότι οι επιστροφές θα πρέπει να είναι ασφαλείς, αξιοπρεπείς και να μην παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Πρόεδρος, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε το λόγο για δύο λεπτά στην ΕΚΟ, γιατί έχουμε και άλλα δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη και πρέπει να δώσουμε το λόγο στον ΕΚΟ. ευχαριστώ πολύ. Όπως ε, υπόθηκε, οι τελευταίες εξελίξεις στην βορειοανατολική Συρία έχουν ε, αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρωπική κατάσταση. Θέλω να πω ε, δύο πράγματα σε σχέση με το τι συνέβη πριν από τον Οκτώβρη και μετά τον Οκτώβρη. Μέχρι τον Οκτώβρη ε, η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ παρήχε ε, περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ ανθρωπιστική και αναπτυξική βοήθεια ε, κατά, κάθε μήνα μέσω προσωπικού που, και ανθρώπων που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή. βασικός στόχος ήταν να, να, να παρέχονται υπηρεσίες διατήρησης της ζωής και μετά τον Οκτώβριο βεβαίω η, κατάσταση, η ανθρωπιστική κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Ε, μιλάμε για εκτοπισμούς και για ε, βάσανα των ανθρώπων που υποφέρουν εδώ και χρόνια λόγω της σύγκρουσης. Θέλω να σταθώ σε δύο σημεία, τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί. Πρώτον, οι οργανώσεις εταίροι μας έχουν παράσχει τεράστια βοήθεια και αρρωγή και δεν έχουν αποχωρήσει από την ε, περιοχή αυτή. Πολλοί διεθνείς εργαζόμενοι έχουν αποχωρήσει, αλλά ε, οι εταίροι μας βρίσκονται ακόμη εκεί. Δεύτερον, το γεγονός ότι η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ ε, παρέσχε την ε, ανθρωπιστική βοήθεια με τον εθελοντικό αυτόν τρόπο, μέσω των εθελοντικών οργανώσεων, αποτέλεσε ζωτική σημασία στοιχείο της βοήθειας που παρήχαμε. Τρίτον, η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι το πώ θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι οργανώσει που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια θα μπορέσουν να συνεχίσουν να το κάνουν αυτό. Διότι η κατάσταση αυτή ε, που έχει διαμορφωθεί ε, επιδεινώνει ε, και μάλλον ενισχύει τις ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι εκεί. Άρα η απάντηση δεν μπορεί να είναι να δοθεί τεθούν λιγότερα στι οργανώσει αυτέ, ούτε να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή των εργαζομένων αυτών των οργανώσεων, διότι δυστυχώ αυτό θα έχει σοβαρέ επιπτώσει και στου πληθυσμού του οποίου θέλουμε να βοηθήσουμε. Και τέλο, η συνέχιση των υπηρεσιών αυτών είναι ζωτική σημασία και εμεί. Να σας πω ότι έχουμε δώσει ανθρωπιστική βοήθεια άνω των 38 εκατομμύριων ευρώ. Το βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας και γι' αυτό το σκοπό θα χρειαστούν να αξιοποιήσουμε όλους τους δρόμους και όλους τους τρόπους ώστε να μπορέσουν εκείνοι που έχουν ανάγκη πραγματικά να λάβουν την βοήθεια που αποστέλουμε εμείς από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την κυρία Αρένα για το ότι μου δίνει δυνατότητα να κάνω κάποιες καταληκτικές ε, ε, παρατηρήσεις πολύ σύντομα, γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση αυτή. Είναι σημαντικό να γίνεται πολιτική συζήτηση, αλλά βεβαίως ακόμα πιο σημαντικό είναι να, να αναλαμβάνονται και δράσεις. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που παρέστησαν σήμερα εδώ στη συνεδρίαση. Θέλω να ευχαριστήσω τους προξεγγλημένους μας Ελπίζω ότι και στο μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα να ε, διεξάγουμε τέτοιες συζητήσεις ε, ανάμεσα στις επιτροπές ΔΕΒΕ και ΝΤΡΟΑ. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους ήρθαν και πάμε τώρα κατευθείαν στο 6 χωρίς ε, διακοπή και σας ευχαριστούμε που περιμένατε. Sorry. Try to make it as short as possible. Alors voilà, on va aborder notre dernier point. Πάμε τώρα στο τελευταίο μας ε, θέμα που είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Αλή Μπιν Σαμίχ. Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κατάρ. Έχουμε πραγματικά υπερβεί τα χρονικά πλαίσια τη ε, συνεδρίαση. οπότε παρακαλώ καθίστε γρήγορα. Αλλά, αλλά, του δίνω τώρα ε, αμέσω το λόγο για να μπορούμε να κάνουμε αυτή την ε, ανταλλαγή και να είναι αυτή όσο παραγωγική γίνεται. Έχετε το λόγο. First Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε την δυνατότητα να σας μιλήσω για τις προόδους και τις ε, δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, πρόκειται για μια καλή ευκαιρία να ανταλλάξουμε μαζί σας πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που έχουμε πετύχει και να ανταλλάξουμε πληροφορίες πάνω στο θέμα αυτό. Θα ήθελα σύντομα να σας ενημερώσω για την Επιτροπή μας, ε, την οποία ιδρύσαμε το 2002. Ε, στο πλαίσιο του Γκάνρι, που είναι ε, η Διεθνής Συμμαχία για την Πρόθεση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Είμαστε ένας από πολλούς οργανισμούς που δημιουργηθήκαμε στο πλαίσιο του σχετικού νόμου. Στόχος μας είναι λοιπόν να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν ξεκινήσαμε τις εργασίες μας το 2002, αντιμετωπίσαμε διάφορες ε, προκλήσεις ε, στη χώρα μας. Πιθανότατα να γνωρίζετε ότι έχουμε υψηλό ποσοστό ε, ε, μεταναστών εργατών οι οποίοι αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για όλες τις στοιχείες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για παράδειγμα τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών. Από τον Ιούνιο του 2017 και μετά αντιμετωπίζουμε νέα προβλήματα μετά τον αποκλεισμό από τις γειτονικές μας χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω σχετικά με τις ε, σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργάτες ε, ε, μετανάστες. Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στο σύστημα Καβάλα, το οποίο στο παρελθόν Ε, υπαγόρευε ότι κανένας ε, μετανάστης εργαζόμενος δεν μπορεί να αλλάξει θέση χωρίς ε, την έγκριση του εργοδότη του. Άλλο θέμα ήταν ότι δεν μπορούσαν να ε, αποχωρήσουν από τη χώρα χωρίς άδεια και έχουν αναφερθεί και τα ψευδή συμβόλαια. Έχουμε μετανάστες από την Ασία, την ε, Ινδονησία, τις Φιλιππίνες, οι οποίοι ε, έρχονται με συμβόλαιο της ε, εταιρείας πρόσληψής τους στη χώρα τους. Ε, καταφθάνουν στο Κατάρ και διαπιστώνουν ότι η σύμβασή τους δεν είναι η ίδια με αυτήν που υπογράψαν στη χώρα τους. Επίσης, έχουμε εμπορία ανθρώπων. Αυτές οι εταιρείε προσλήψεων ε, απλά θέλουν να πάρουν τα χρήματα των μεταναστών. Άλλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί στη χώρα μας ε, σχετίζεται με την καθυστέρηση καταβολής των μισθών τους. Ξεκινήσαμε το 2004 με υποβολή συστάσεων στην κυβέρνησή μας ε, να καταργήσει το σύστημα Καβάλα. Το 2009 είχαμε ε, κάποια πρόοδο. Ε, το 2009 όμως δεν άλλαξε σημαντικά ο νόμος μετά από το Μοντιάλ το 2010 ε, πραγματοποιήθηκε μια ευρεία εκστρατεία. Ως ε, Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήμασταν ικανοποιημένοι με την εκστρατεία αυτή και τις ε, συστάσεις προς την κυβέρνησή μας και από πλευράς του, της, της ITUC. Ιδιαίτερα από το 2013 και μετά, έχουν σημειωθεί πρόοδοι και το σημαντικότερο όσον αφορά το σύστημα αυτό είναι ότι άλλαξε η νομοθεσία το 2015. Πριν την αλλαγή της νομοθεσίας δεν μπορούσε κανείς να αλλάξει η θέση εργασίας χωρίς την ε, ε, συγκατάθεση του εργοδότη του. Τώρα όμως μπορεί πια με βάση τη σύμβαση που έχει υπογράψει με την ε, επιχείρηση ή με τον εργοδότη του. Επίσης τροποποιήθηκε το άρθρο υπαριθμών 7 του νόμου το 2015. Και καταργήθηκε η άδεια εξόδου από τη χώρα. Έτσι, το 90% των μεταναστών μπορούν τώρα πια να εξέλθουν από τη χώρα χωρίς την άδεια του εργοδότη τους. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το σύστημα αυτό. Όταν μιλάμε για τις ε, συμβάσεις ή ψευδείς ε, συμβάσεις, υπάρχουν κάποιες ε, συστάσεις από την διεθνή κοινότητα. Ζητήσαμε από την κυβέρνησή μας να λύσει το πρόβλημα, ώστε προτού καταφτάσουν μετανάστες στη χώρα μας, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στη χώρα τους διότι οι ε, εταιρείε πρόσληψης ε, παίρνουν τα χρήματά τους ε, και τους δίνουν ψευδή συμβόλαια. Τώρα λοιπόν έχει δημιουργηθεί σύστημα το οποίο εφαρμόζεται με 8 χώρες της Ασίας, το Μπαγκλαντές, την Ινδία και άλλες χώρες. Υπάρχουν λοιπόν κέντρα έκδοση θεωρήσεων. Έτσι λοιπόν πριν καταφτάσουν οι άνθρωποι αυτοί στο Κατάρ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πρόκειται για σύμβαση που υπογράφεται πριν καταφτάσει και λαμβάνει τη σύμβαση στη γλώσσα του εργαζόμενος, έτσι γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του. όσον αφορά τις ε, καθυστερήσεις στην καταβολή των ε, μισθών. Το 2014 η κυβέρνηση δημιούργησε μια ρύθμιση προστατευτική Παλαιότερα λάμβανε σε μετρητά ο εργαζόμενος τα χρήματά του. Με την αλλαγή αυτή όμως παρακολουθείται η καταβολή των ε, μισθών, διότι γίνονται πια μέσω των τραπεζών. Έτσι το Υπουργείο Εργασίας παρακολουθεί τις ε, μεταφορές των χρημάτων. Επίσης ε, δημιουργήθηκε η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Κατόπιν, το 2018 εκδόθηκε νέα νομοθεσία που ε, παρέχει διασφαλίσεις για τους ε, μετανάστες εργαζομένους. Πολλοί από αυτούς σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας τη επιχείρηση ε, δεν ε, λάμβαναν τα χρήματά τους. Τώρα πια όμως υπάρχει αυτό το ταμείο το οποίο ε, καταβάλει τους μισθού των ανθρώπων αυτών και κατόπιν τους ζητάει από την ίδια την επιχείρηση. Υπάρχουν επίσης νομοσχέδια σχετικά με τον ελάχιστο μισθό. Το Υπουργικό Συμβούλιο συμφώνησε πάνω στη σχετική νομοθεσία τον προηγούμενο μήνα. Αυτές λοιπόν είναι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει. Η κυβέρνησή μας ε, λοιπόν έτσι αντιμετωπίζει τα προβλήματα που είχαμε με εργαζόμενους μετανάστες. Εμείς όμως ως Οργανισμός ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πιστεύουμε ότι ε, είχαμε προκλήσεις, υποβλήθηκαν συστάσεις. Η βασική πρόκληση τώρα όμως είναι πώς θα εφαρμόσουμε στην πράξη όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις, ε, διότι είχαμε πολλές προκλήσεις ε, πριν ξεκινήσουν οι μεταρρυθμίσεις. Τώρα έχει υπογραφεί συμφωνία με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το ILO. Ο ILO υποστηρίζει το Υπουργείο Εργασίας ε, στην εφαρμογή όλων των μεταρρυθμίσεων. Τον προηγούμενο μήνα, το γραφείο του ILO στην Ντόχα εξέδωσε έκθεση προόδου σχετικά με την ε, επίλυση όλων των προβλημάτων. Αυτή λοιπόν είναι η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Από τον Ιούνιο του 2017 και μετά αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις. Ξεκίνησε η κρίση του κόλπου τον Ιούνιο του 2017 και ε, τα Ηνωμένα Αραβικά ημεράτα το Μπαχρέιν, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία ε, απέκλεισαν το Κατάρ. Αυτή βέβαια είναι μια κυρίαρχη απόφαση από πλευράς κάθε κράτους. Από την άλλη πλευρά όμως ε, εφήρμοσαν καταναγκαστικά μέτρα εις βάρος των ανθρώπων. Πρόκειται για συλλογική τιμωρία, ε, κατά τη γνώμη μας. Ε, πρόκειται για διαχωρισμό οικογενειών. Ε, απέβαλαν όλους τους φοιτητέ από τις χώρες τους. Ζήτησαν από τους υπηκόους μας να... ζήτησαν από τους υπηκόους τους να εγκαταλείψουν το Κατάρ μέσα σε δύο εβδομάδες χωρίς να λάβουν καθόλου υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Εμείς ε, εκδώσαμε ε, μια δήλωση και πολλές εκθέσεις ε, σχετικά με το θέμα αυτό και ζητήσαμε από τον είπα το Επίτροπο να εξετάσει εάν είναι νόμιμα όλα αυτά τα καταναγκαστικά μέτρα. Είχαμε μια τεχνική αποστολή που εκπώνησε έκθεση όπου μιλάει για συλλογική τιμωρία των ανθρώπων αυτών και καταναγκαστικά μέτρα. Ζήτησε λοιπόν από όλες τις χώρες αυτές να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους. Από την άλλη υπάρχουν και πολλές εκθέσεις της διεθνούς κοινότητας. Είδαμε έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, ε, της Human Rights Watch και η κυβέρνησή μας προσέφυγε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ζητώντας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να αναθεωρήσουν την απόφασή τους. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ζήτησε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να επιτρέψουν επανένωση των οικογενειών και να επιτρέψουν και επιστροφή των φοιτητών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Δυστυχώς η διερμηνής θα είναι μαζί μας μέχρι τις 6.30 μόνο και ξέρω ότι κάποια μέλη της Επιτροπής μας δυσκολεύονται αν δεν υπάρχει διερμηνία, γι' αυτό και... Άρα είσαι η πρόεδρος της αντιπροσωπείας ε, και ξέρω λοιπόν ότι, ότι θα έχει πρόβλημα να έχουμε δερμηνία, όχι δεν σε πειράζει. Καλά, τότε να μυρίζει πρώτα η Άννα και μετά εσύ συνάδελφα. Ευχαριστώ. Έχουμε ξανασυναντηθεί. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω κύριε Ζαμάρη εδώ στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θέλω να ε, σα συγχαρώ εσά και την οργάνωσή σα που έχετε λάβει πλέον ε, και το καθεστώς ε, οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολα. Εγώ ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να προστατεύονται και να διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη την Αραβική Χερσόνησο, όχι μόνο στο Κατάρ. Γι' αυτό και θα προσκαλέσουμε στην Επιτροπή και άλλους ε, αξιωματούχους της περιοχής, ε, ανθρώπους από την περιοχή. Ε, πάντως, θέλουμε πραγματικά η οργάνωσή σας να είναι εταίρος μας, δεδομένου ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κατάρ εξακολουθεί να είναι προβληματική και θα μου επιτρέψετε να κάνω κάποιες ερωτήσεις ως προς αυτό. Δικαιώματα των γυναικών. Θα ήθελα να μου πείτε τι κάνει η δική σας οργάνωση όσον αφορά την, ε, τα δικαιώματα των γυναικών και την εναπομείνασα ε, νομοθεσία που κάνει διακρίσεις βάρος των γυναικών, ιδίως όσον αφορά την κυδαιμονία των παιδιών και τα κληρονομικά θέματα. Επίσης, πολλές γυναίκες έχουν προβλήματα ε, να εγγραφούν και να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στο Κατάρ. Είπατε επίσης ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδο όσον αφορά του μετανάστε στο Κατάρ. Είπατε επίσης ότι το 90% των εργαζομένων έχουν ε, πλέον την ελευθερία να εγκαταλείψουν τη χώρα ε, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Το άλλο 10% επίσης. Είπατε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά. Το ερώτημά μου όμως είναι, γίνονται έρευνες για τα εκατοντάδες θύματα, τους εκατοντάδες θανάτους που είχαμε τα τελευταία χρόνια, εργαζομένων, λόγω της ε, ε ζέστης που επικρατεί στη χώρα. Τα εργατικά αυτά ατυχήματα και το γεγονό ότι η λήψη προληπτικών μέτρων είναι απλά εθελοντική από τις επιχειρήσεις. Και θέλω να σας απευθύνω και ένα ερώτημα σχετικά με το εμπάργο που έχει επιβληθεί στο Κατάρ. Στην έκθεση 2018 είπατε ότι είχατε 4.000 καταγγελίες όσον αφορά το εμπάργο και 1.800 καταγγελίες ε, που αφορούσαν Άλλε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορείτε να μα πείτε ε, τι αφορούσαν αυτέ οι άλλε οι 1800 άλλε καταγγελίε. Ευχαριστώ ο κύριο Ταραμπέλα ω αντιπρόεδρο τη αντιπροσωπεία. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Μου δώσετε αυτά δύο λεπτά και θα τα εκμεταλλευτώ και σα ευχαριστώ κύριε πρόεδρε για την ομιλία σας όσον αφορά τα δικαιώματα των ε, μεταναστών ε, εργαζομένων. Τα έχουμε πει αυτά με το Intergroup για τον αθλητισμό, μιλήσαμε και για το κατάλληλο στο παρελθόν και βέβαια μας απασχολούν τώρα όλα αυτά γιατί ασχολούμαι ακόμη με τις ε, χώρες και τις περιοχές και μπράβο μας είπατε για την πρόοδο που σημειώσατε ε, να μην επαναλάβω τα επιτεύγματά σας. Υπάρχει επομένως αυτή η εξέλιξη. Ε, ξέρουν τι πρέπει οι αρχές της χώρας για τους εργαζομένους. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή η θετική τάση θα συνεχιστεί. Ε, γιατί φυσικά απομένουν ακόμα πολλά πρέπει να γίνουν στο μέλλον. Επίσης όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο του 22, ε, είδατε τι έγινε τον Δεκέμβριο, είχαμε όλες αυτές τις ε, τα θέματα σε σχέση με το ότι θα κάνει πάρα πολύ ζεστή εκεί. Ε, ε, βέβαια και αυτοί που διαμαρτύρονται, Αργεντινή, Βραζιλία, ε, εντάξει και αυτοί έχουν συνηθίσει το, τη ζέστη. Τώρα για πέστε μας εσείς, για το περιβάλλον τι θα κάνετε όσον αφορά το, το να φτιάξετε τέτοιες υποδομές γιατί ε, άλλωστε σήμερα δεν μπορούμε να μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τη, την θέρμα, αναθέρμανση πάντων του πλανήτη, ε, υπερθέρμανση μάλλον, γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα που θα αφορά το αποτύπωμα του άνθρακα. Και τώρα ε, διακόπτουμε λεπρόδος και ευχαριστούμε για την ερμηνεία λεπρόδος και εμείς. <laughs> We're all free to let